Καθίστε παρακαλώ όλες και όλοι και τότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε και καθώς ε, θα λαμβάνετε τις θέσεις σας, θα κάθεστε. Θα ήθελα να παρακαλέσω να εγκρίνουμε την ημερεσία διάταξη και επιτρέψτε μου να αναβάλω τις ανακοινώσεις της Προέδρου για αύριο, ώστε να μην φάμε το χρόνο που διαθέτουμε για τη συζήτηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν συμφωνείτε λοιπόν, δεν βλέπω να ε, ενίσταται κανείς. Έχουμε επίση πολλά πρακτικά συνεδριάσεων τα οποία πρέπει να εγκριθούν. Μπορώ να τα διαβάσω και απευθείας από την ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια πρακτικών έχουν περιληφθεί σε μεγάλο βαθμό μόνο στα αγγλικά και επειδή είναι η τελευταία μας συνεδρίαση του έτους, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να περιλάβουμε στην σημερινή ημερήσια διάταξη τα εκκρεμή πρακτικά, όσο δυνατόν περισσότερα δηλαδή από τα εκκρεμή πρακτικά του 2012. Και σημειώστε ότι τα υπόλοιπες γλώσσες των πρακτικών θα είναι διαθέσιμες οι μεταφράσεις δηλαδή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Λοιπόν, έχουμε τώρα 2 Ιουλίου, 10 Σεπτεμβρίου, 24 και 26 Σεπτεμβρίου, 10, 15 και 22 Οκτωβρίου 2012, 12 Νοεμβρίου, 15 Νοεμβρίου και 19 Νοεμβρίου 2012. Αυτά τα πρακτικά λοιπόν παρακαλώ να εγκρίνετε. Προφανώς τα έχετε λάβει όλοι. Ουδής ενίσταται. Πολύ καλά αφήνω τις ανακοινώσεις της Προέδρου που όπως είπα θα τις ε, ακούσετε αύριο και με μεγάλη χαρά καλωσορίζω ακόμη μια φορά τον κύριο Ντράγκη εδώ στην Επιτροπή μας, είναι συχνός επισκέπτης μας. Θα κάνει εισαγωγικές παρατηρήσεις της τάξης των 10 λεπτών, θα ακολουθήσει ένας γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων και θα ακολουθήσουμε τον νέο αυτό τρόπο που έχουμε αποφασίσει, δηλαδή 5 λεπτά για κάθε ε, ε, ερώτηση και απάντηση. Αν σας μείνει κάποιος χρόνος, μπορείτε να ξαναλάβετε το λόγο. Αν όμως μείνετε στα πέντε λεπτά με την ερώτησή σας τα 30 τελευταία δευτερόλεπτα, τότε θα προλάβετε να την κάνετε. Πάντως καλά τα καταφέραμε τις άλλες φορές όταν ε, διεξαγάγαμε τις ακροάσεις των επιτρόπων και κάποιους άλλους οικονομικούς διαλόγους. Γι' αυτό ας προχωρήσουμε τώρα στον νομισματικό διάλογο να δούμε εάν ίσως μπορούμε να αντλήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τον κύριο Ντράγκη γιατί λίγο πολύ αυτός είναι ο στόχος μας. Μάριο θα σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι πάλι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενώπιόν σας για την τελευταία ανταλλαγή απόψεων του 2012. Φέτος, ο χρόνος αυτός δεν ήταν εύκολος. Δοκιμάστηκαν οι δεσμοί των χωρών μελών, κυρίως της Ευρωζώνης. Ωστόσο, αναπτύχθηκε και ένα μακροοικονομικό όραμα της ε, Ευρωζώνης και είναι ένα έτος όπου αυτό το όραμα άρχισε να μεταφράζεται σε δράσεις και για σημαντικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Τελειώνουμε τον χρόνο με θετική νότα, ξεκινώντας αυτό το μακροπρόθεσμο όραμα με τα ενεργά βήματα που λαμβάνουν και κυβερνήσεις και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προς την κατεύθυνση μιας αληθινής Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και πιο ε, πρόσφατα ακόμη με την ομόφωνη απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ να δημιουργήσει το ενιαίο ε, μηχανισμό εποπτείας. Συγχαίρω την Επιτροπή σας για την ταχεία υιοθέτηση της θέσεώς της για αυτόν ακριβώς τον μηχανισμό και για την φιλόδοξη ευρωπαϊκή της προσέγγιση. Πρόκειται για ξεκάθαρη απόδειξη ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι αποφασισμένα να δράσουν με τρόπο ε, έγκαιρο και αποφασιστικό, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Είναι επίση μια σαφή ένδειξη για το γεγονό ότι οι χώρες μέλη της ζώνης ευρώ είναι έτοιμε να συμφωνήσουν πάνω σε μια ε, σημαντική, ε, σε ένα σημαντικό μοίρασμα της κυριαρχίας εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις έχουν γίνει βήματα προς μια σταθερότερη Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Η δημιουργία του μηχανισμού SSM, ενέα εποπτείας δηλαδή, θα αποτελέσει ένα κέριο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ο μηχανισμός SSM θα συνεχίσει να εμπνέει εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα σε όλη τη ζώνη ευρώ. Θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση των ε, δανειοδοτήσεων μεταξύ τραπεζών και των ροών των πιστώσεων διασυνοριακά και σε συνδυασμό με την απευθείας ανακεφαλαίωση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, καθώς και με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, αυτός θα επιτρέψει να ξεπεραστούν ε, οι δυσκολίες μεταξύ δημοσίου χρέους και τραπεζών. Ελπίζω ότι η νομισματική ε, διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα. Μετά από την έγκριση των σχετικών νομικών πράξεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ξεκινήσει τις προετοιμασίες έτσι ώστε ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας να μπορέσει να καθιδρυθεί μέσα στα χρονικά όρια που έχουν προβλέψει οι νομοθέτες. Στις σημερινές μου εισαγωγικές παρατηρήσεις θα σας δώσω πρώτα μια σύντομη εποπτεία της οικονομικής και νομισματικής καταστάσεως και μετά θα έλθω στην σχέση μεταξύ νομισματικής πολιτικής και οικονομικής εποπτείας, δημοσιονομικής εποπτείας. Και θα κλείσω εξηγώντας τις απόψεις μου για τις προτεραιότητες για το 2013, για την εφαρμογή δηλαδή αυτού του κοινού μακροπρόθεσμου οράματος για την Ευρωπαϊκή ε, Νομισματική Ένωση. Μετά από την τελευταία μας συνάντηση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφησε απαράλλαχτα τα βασικά της επιτόκια το βασικό αναχρηματοδότησης είναι στο 0,75%. Για την deposit facility έχει παραμείνει στο μηδενικό και για την marginal lending έχει στο 1,5%. Για άλλα μέτρα που δεν είναι στάνταρ της νομισματικής πολιτικής, το Συμβούλιο μας αποφάσισε τον Δεκέμβριο να συνεχίσει να διεξάγει όλες τις επιχειρήσεις αναχρηματοδότησης με ε, σταθερό επιτάκιο, επιτόκιο μέχρι τουλάχιστον τον Ιούλιο του 2013. Μεσοπρόθεσμα η οικονομική δραστηριότητα παραμένει πρόκληση. Για, τρίτο, για δεύτερο μάλλον συνολικό τρίμηνο και οι ενδείξεις για το τέταρτο τρίμηνο δείχνουν σημαντικές αδυναμίες παρόλο που ορισμένοι πρόσφατοι δείκτες έχουν σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα και η ψυχολογική κατάσταση της οικονομικής αγοράς έχει βελτιωθεί κι άλλο. Η εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να είναι χαμηλή λόγω της ψυχολογίας και των επενδυτών και των καταναλωτών καθώς και των, του τραπεζικού τομέα που ακόμα αναμένει τις αποφάσεις για τις επενδύσεις. Αναμένουμε η οικονομική αυτή αδυναμία να συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο με πολύ σταδιακή ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους. Η ανάκαμψη αυτή αναμένεται να στηριχτεί από την ενίσχυση της παγκόσμιας ζήτησης, από την ε, νομισματική πολιτική, καθώς και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις οικονομικές αγορές, που θα πρέπει να καταλήξουν και σε αποφάσεις για επενδύσεις και δαπάνες. Έχει συνεχίσει ο πληθωρισμός να παραμένει μέτριος. Από το 2,5% τον Οκτώβριο έφτασε το 2,2% τον Νοέμβριο. Αναμένεται να μειωθεί κι άλλο στο μέλλον. Και αυτό θα ενισχύσει τα πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα. Για την, ε, για την ανάπτυξη των τιμών Αυτές αναμένονται να παραμείνουν μέσα στα πλαίσια των στόχων του Διοικητικού μας Συμβουλίου και κάτω από 2% αλλά κοντά στο 2%. Η νομισματική μας ανάλυση μας δίνει μια εικόνα που είναι συνεπής με τη σταθερότητα των τιμών. Εξετάζοντας τις εξελίξεις για πολλούς μήνες, η νομισματική επέκταση, εφόσον λαμβάνει υπόψη και συγκεκριμένους ε, παράγοντες, παραμένει χαμηλή. Οι δυναμικές των, ε, των, ε, των δανείων επίσης είναι χαμηλές και σε πολλά μέρη της Ευρωζώνης έχουν συρρυκνωθεί. Και αυτό οφείλεται στις προσαρμογές των ισολογισμών, των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Το πρώτο θέμα τώρα που έχουμε διαλέξει για την ανταλλαγή απόψεών μας, που είναι η σχέση μεταξύ νομισματικής πολιτικής και δημοσιονομικής εποπτείας. Οι συζητήσεις που οδήγησαν στην πρόσφατη απόφαση για την καθίδρυση του εποπτικού μηχανισμού έχουν θέσει και το ερώτημα με ποιον τρόπο θα πρέπει να διαχωριστούν οι πολιτικές οι νομισματικές πολιτικές από τις ευθύνες για την εποπτεία. Τα τελευταία χρόνια πολλές κεντρικές τράπεζες για τους δικούς τους σωστούς λόγους έχουν αναλάβει εποπτικό ρόλο. 14 από τις 17 εθνικές κεντρικές τράπεζες στην ζώνη ευρώ παίζουν ρόλο στην εποπτεία. Το ίδιο πράττουν πολλές κεντρικές τράπεζες και αλλού στον κόσμο. Πράγματι, η παγκόσμια οικονομική κρίση οδήγησε σε στενότερους δεσμούς μεταξύ κεντρικών τραπεζών και της δημοσιονομικής εποπτείας. Η Τράπεζα της Αγγλίας, για παράδειγμα, σύντομα θα αναλάβει εποπτικές ευθύνες που προηγουμένως είχε αναλάβει η Financial Services Authority. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τον ρόλο του Fed στην δημοσιονομική εποπτεία τον έχουν ενισχύσει. Όλα αυτά δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ νομισματικής πολιτικής και δημοσιονομικής εποπτείας παίζει σημαντικό ρόλο ιδίως σε περίοδους κρίσεως. Δεν είναι και τυχαίο που ιστορικά οι πρώτες κεντρικές τράπεζες ήταν επόπτες, είχαν την εποπτεία, επί των εμπορικών τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εκδώσει ξεκάθαρες κατευθύνουσες αρχές και εσωτερικές ε, πρακτικές για να επιτύχει την αποτελεσματικ... τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των δύο πολιτικών, δηλαδή της νομισματικής πολιτικής και της εποπτείας. Πρώτα, η εμπλοκή της στην δημοσιονομική εποπτεία δεν έχει απολύτως κανένα αποτέλεσμα επί του βασικού μου στόχου που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Ούτε επί του στόχου, που αυτός είναι δεσμευτικός νομικά, ούτε και από την ποσοτικοποιημένη έκφραση σε ε, ρυθμό πληθωρισμού που είναι περίπου στο 2%. Δεύτερο, ένα supervisory board, εποπτικό συμβούλιο, θα αποτελεί το κέντρο για τη διαχείριση και την, της, εποπτικής, ε, της ε, δημοσιονομικής εποπτείας. Με γεωγραφική ενότητα που θα είναι κάπως ευρύτερη από τη ζώνη ευρώ, εφόσον, όπως ελπίζουμε, ορισμένες χώρες οι οποίες επί του παρόντος δεν είναι μέλη της ζώνης ευρώ, ωστόσο θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στον εποπτικό μηχανισμό. Τρίτο, ο χωρισμός μεταξύ νομισματικής πολιτικής και ε, δημοσιονομικής εποπτείας θα λάβει ιδίω την μορφή ανεξάρτητης ανάλυσης και υποβολής συστάσεων για την χρήση των εργαλείων πολιτικής και για τις δύο αυτές λειτουργίες. Αυτό θα βασίζεται σε μια ισχυρή διακυβέρνηση. Εμείς θα καθιερώσουμε από τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες θα διασφαλίσουν την το ξεκάθαρο αυτό διαχωρισμό ακολουθώντας τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. Ο διαχωρισμός των δύο λειτουργιών είναι ουσιώδης. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η ισχυρότερη εποπτεία διευκολύνει και την διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής. Εδώ δύο παράδειγματα. Πρώτα, απουσία δημοσιονομικής σταθερότητας τα στάνταρ εργαλεία της νομισματικής πολιτικής, δηλαδή αλλαγές των επιτοκίων, χάνουν κάποια από την ισχύ τους. Η αποτελεσματική εποπτεία που συμβάλλει στη σταθερότητα των δημοσιονομικών συστημάτων δεν μπορεί παρά να ωφεληθεί από την ομαλή μεταβίβαση της νομισματικής πολιτικής. Δεύτερο, η αποτελεσματική δημοσιονομική εποπτεία μπορεί να αποτελέσει το αντίβαρο στο υπερβολικό, στην υπερβολική μόχλευση και τις επεκτάσεις πιστώσεων. Έτσι, μειώνοντας τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, η αποτελεσματική εποπτεία μπορεί να σφυριλατήσει ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον με σταθερές τιμές. Η νομισματική πολιτική θα παραμείνει προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της σταθερότητας των τιμών ώστε να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των αγορών και του κοινού για την αγοραστική, αξία, του, αγοραστική δύναμη του νομίσματος. Αυτό μειώνει την επιτητικότητα και δημιουργεί ένα περιβάλλον σταθερών ε, οικονομικών αγορών. Αρχίσαμε ήδη με τον εσωτερικό προβληματισμό για όλα τα θέματα αυτά, μαζί με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και τυπικά τις προετοιμασίες μόλις θα είναι έτοιμο το απαραίτητο νομικό πλαίσιο. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα που έχουμε επιλέξει για την ανταλλαγή απόψεών μας σήμερα, δηλαδή μια γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση. Την άνοιξη φέτος, μετά από τρία χρόνια σημαντικών οικονομικών και δημοσιονομικών προκλήσεων, κατέστη σαφές ότι αυτό που χρειάζεται η ζώνη ευρώ είναι ένα συνεκτικό μακροπρόθεσμο όραμα για μια οικονομική για μια Ευρωπαϊκή συγγνώμη, Νομισματική Ένωση. Στην ακρόαση του Απριλίου συζητήσαμε το όραμα αυτό μετά από προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε κάνει στην παρούσα Επιτροπή για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και για το Σύμφωνο ανάπτυξη. Το όραμα που είχε καταστροφεί τότε με μεγάλη λεπτομέρεια από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Από τότε έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου απετέλεσε σημαντικό ορόσημο. Θεσμικές αλλαγές που ήταν αδιανόητες μόλις πριν από ένα χρόνο, βρέθηκαν τώρα στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρόκειται να λάβουν τελική μορφή. Ο μηχανισμός εποπτείας είναι ένα κύριο παράδειγμα αυτής της πολιτικής φοράς. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε και άλλα βήματα για την ολοκλήρωση του μηχανισμού εποπτείας. Οι συζητήσεις σε βάθος για μεταρρυθμίσεις και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας δηλαδή, έπαιξαν σημαντικό ρόλο και απηχούνται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Από την οπτική γωνιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εγώ βλέπω δύο βασικές προτεραιότητες για το 2013. Πρώτα, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Οικονομικής Ένωσης. Οι υπερβολικές ανισορροπίες μέσα στην ίδια την ε, ζώνη ευρώ έχουν αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά. Μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι φαίνεται καθαρά τώρα να αρχίζει μια προσαρμογή. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έχουν αυξηθεί κατά 27% κατά όγκων στην Ισπανία από το 2009, 14% στην Ιρλανδία, 22% για την Πορτογαλία και 21% για την Ιταλία. Οι τέσσερις αυτές χώρες σημειώνουν επίσης κέρδη και στο συγκριτικό κόστος μονάδας εργασίας. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, έστω και αν βραχυπρόθεσμα το κόστος για τους επιμέρους πολίτες είναι και μπορεί να είναι και είναι πραγματικά πολύ βαρύ. Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις είναι ωστόσο δρόμος και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιμείνουν στον δρόμο αυτό. Τι μπορεί να γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να δοθεί ακόμα περισσότερη υποστήριξη στην διαδικασία αυτή. Οι προτινόμενες συμβάσεις ε, μεταρρυθμίσεων, reform contracts μεταξύ χωρών μελών της Ζώνης Ευρώ και των ε, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόσχονται πολλά και συνδυασμένε με ένα πλαίσιο στοχευμένης και προσωρινής υποστήριξης θα μπορέσουν να σφυριλατήσουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές Αλλαγέ και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα reform contract θα πρέπει να στοχεύσουν ιδίω σε χώρες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερε προκλήσεις ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να εντοπίσουν τις διαφορετικές εχμές για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και να στοχεύσουν καλύτερα τις μεταρρυθμίσεις. Κάτι το οποίο θα καθιερώσει ένα, ένα, ε, μια διασύνδεση μεταξύ των μεταρρυθμίσεων και της ανταγωνιστικότητας που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η λειτουργία των αγορών προϊόντων και εργασίας είναι απαραίτητη για να υπάρξει ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Γι' αυτό χαίρομαι για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τον επόμενο χρόνο θα προχωρήσει σε συστηματική επανεξέταση των αγορών αγαθών και εργασίας. Για τις χώρες της ζώνης ευρώ η ε, επιθεώρηση αυτή θα πρέπει να επιτρέψει να εκτιμηθεί εάν οι αγορές αυτές συμβαδίζουν απολύτως με τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Εδώ οι αγορές αγαθών και εργασίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον το οποίο αλλάζει και να μπορούν να διατηρήσουν και ψηλά επίπεδα απασχόλησης. Η δεύτερη προτεραιότητα για το 2013 από την σκοπιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η ολοκλήρωση της Δημοσιονομικής Ένωσης με την καθιέρωση ενός ενίου μηχανισμού επιλύσεων. Διαλύσεως ή εξαγοράς τραπεζών διορθών. Που αυτός είναι σημαντικός στόχος και θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε και την δημοσιονομική σταθερότητα. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέψει στις τράπεζες να πτωχεύουν με τρόπο τακτικό, όχι άτακτο δηλαδή. Περαιτέρω βελτίωση της Οικονομικής Ένωσης με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και με, και με ένα ενιαίο πλαίσιο από την άλλη μεριά είναι βασικές μας προτεραιότητες για το 2013. Η παρούσα Επιτροπή πάντοτε πρόσφερε όθηση για φιλόδοξες ευρωπαϊκές λύσεις στον τομέα της δημοσιονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης και είμαι πεισμένο ότι και πάλι θα παίξετε ένα κέριο ρόλο για να προχωρήσει η ατζέντα αυτή και να εγκριθούν οι απαραίτητε νομοθετικέ προτάσεις. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας και πολύ ευχαρίστω θα απαντήσω στι ερωτήσει σα. we're now going to move to the uh, question and σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δράγη. Ας περάσουμε στην περίοδο των αραταπαντήσεων. Ξέρω ότι ο Μάριο πρέπει να φύγει στις 5.30 ακριβώς, οπότε να είστε σύντομοι. Ε, οι χρονοθυρίδες σας δεν μπορούν να υπερβούν τα 5 λεπτά. Αυτό είναι ο χρόνος που δόθηκε από τους ε, συντονιστές. Εάν λοιπόν μακρηγορείτε, θα χρειαστεί μετά να περιορίσω το χρόνο απάντησης του Προέδρου της ΕΚΤ. Ο, ο Παύλος Ζέλμπα πρώτα. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Πράγματι, ήταν δύσκολη χρονιά, συμφωνώ μαζί σας, ωστόσο έγιναν σημαντικά βήματα. Αναγνωρίσατε ότι με την απουσία δημοσιονομικής σταθερότητα, η νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε. Στην Ισπανία έχουμε προφανείς δείκτε οι οποίοι δείχνουν, δείχνουν ότι τα πράγματα τα κάνουμε σχετικά καλά. Βελτιώνεται και αυξάνεται η παραγωγικότητα, μειώνεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας όπως αναγνωρίσατε και εσείς ο ίδιος. Οι εξαγωγές μας από το 2009 αυξήθηκαν κατά 27%. Συν της οι μεγάλες πολυεθνικές που δεν εξαρτώνται από την πίστοση των Ισπανικών τραπεζών κάνουν πράγματι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας. Το πρόβλημα όμω, κύριε Ντράγκη, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας μας και οι οποίες εξαρτώνται από την πρόσβαση που θα έχουν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει κλείσει τη στρόφιγγα και γι' αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλε δυσκολίε. Δεν μπορούν βεβαίω να δημιουργήσουν θέσεις απασχόληση και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωση. Εξαρτάται λοιπόν η επιβίωση της επιχείρησης από το που έχει την έδρα της γεωγραφικά, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι πλήγμα στην ενιαία αγορά και πλήττει και την παραγωγικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ερωτώ λοιπόν, τι μπορεί να κάνει η νομισματική πολιτική για να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση ή τουλάχιστον, εν περιπτώσει, να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. Όντω, τα πράγματα προχωρούν στην Ισπανία και θα έλεγα και σε όλες τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε όλα τα μέτωπα που αναφέρατε. Επίσης, αληθεύει ότι οι ροές πίστοση παραμένουν περιορισμένες. Το πρώτο τμήμα του έτους με τις, τα δύο προγράμματα δώσαμε περίπου μισό τρει στο σύστημα. Αλλά τα χρήματα αυτά δυσκολεύονται να βρουν το δρόμο τους προς την οικονομία. Υπάρχουν δύο μεγέθη στην ανάπτυξη των πιστώσεων. Η μία είναι η, η παροχή, η προσφορά. Αποφεύγουμε δηλαδή και προστατεύουμε τις τράπεζες που μπορεί να αντιμετωπίσουν ε, ατυχήματα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και έπειτα ε, επεκτείνουμε το παράπλευρο πλαίσιο έτσι ώστε πολλές τράπεζες που πιέζονται όπως στην Ισπανία να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση που προσφέρεται από το από την επιχείρηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Ε, ωστόσο οι τράπεζες παραμένουν ε, επιφυλακτικές και περιορίζεται η ροή πίστοσης. Τι μπορούμε να κάνουμε, να δεχθούμε αυτό που λέγεται επιπλέον απαιτήσει πίστοσης ως παράπλευρη ε, έννοια σε σχέση με τις πιστώσεις που μπορούν να πάρουν από την ΕΚΤ. Εμείς λάβαμε μια πολύ σοβαρή απόφαση. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε αυτή την επιπλέον ρευστότητα και αυτή να μπορέσει να βρει δρόμο, το δρόμο προς την οικονομία. Γιατί η τράπεζες αυτές δανείζονται και μπορούν έτσι να το χρησιμοποιήσουν αυτό ως εγγύηση για να δανειστούν στη συνέχεια από την ΕΚΤ. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δούμε ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο παράγοντας ζήτησης και πώς θα αναπτυχθεί. Ωστόσο, είμαστε βέβαιοι ότι δεδομένη της τάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή η καλή επιρροή θα γίνει αισθητή και στην οικονομία γιατί με βάση τις προβλέψεις της ΕΚΤ βλέπουμε και προβλέπουμε μάλλον μια αρχή ανάκαψης για το δεύτερο ήμιση του έτους. Uh, Ευχαριστώ και τώρα η Ελίζα Φερέιρα από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντράγκη ε, που είστε εδώ μαζί μας. Τα πρώτα μου λόγια είναι για να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστήσουμε γιατί η μακροπρόθεσμη οπτική και όραμα που δώσατε για την, για την Ένωση, την Νομισματική Ένωση, η αντιμετώπιση των κερδοσκόπων, αλλά και τώρα η Τραπεζική Ένωση. Νομίζω πως ε, το ενιαίο νόμισμα θα είχε διαλυθεί αν δεν υπήρχαν αυτές οι παρεμβάσεις. Του του λεχθέντος ε, διαφωνώ με την οπτική που έχετε σε σχέση με το οικονομικό ε, τμήμα, δηλαδή την πραγματική οικονομία και την εξέλιξη της. Γιατί, και, ε, διότι η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση. 25 εκατομμύρια άνεργοι. Το έλλειμμα και το χρέος αυξάνονται και οι χώρες, ε, πολλές χώρες είναι σε υπό συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παρακαλώ κάντε μια απόπειρα με βάση όλα αυτά τα θέματα, λογικό και αντικειμενικό και όχι παράλογο σε σχέση με τα όσα γίνονται. Όταν μια οικονομία ε, στην ουσία έχει καταρρεύσει πρέπει να περιορίσουμε τις δόσεις σε λιτότητα. Αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες που είναι υπό συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στην Πορτογαλία σήμερα ε, έχουμε ενώπιόν μας ένα σημαντικό κίνδυνο αποπληθωρισμού. Και πιστεύω επίσης και θα ήθελα να γνωρίζω αν οι συνθήκες και θα ήθελα να απαντήσετε για τις χώρες που ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν αυτοί οι όροι θα μπορούσαν να μοιραστούν σε όλους. Δηλαδή, μήπως οι τα καλύτερα μέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και από άλλους. Γιατί τα κέρδη τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιστρέφονται στις ε, χώρες με βάση τις οποίες τελικά επετέφθησαν. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε για μένα. Μην ξεχνάμε, το ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και το Σύμφωνο ανάπτυξη για πρώτη φορά ακούστηκαν εδώ, στο Κοινοβούλιο. Και εγώ θα πρέπει να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΕΚΟΝ για τις γόνιμες συζητήσει που βρίσκονται στην πηγή αυτών των δύο ενιών και ιδεών. Και τώρα, ερχόμενο στην ερώτησή σας, θα ήθελα να πω ότι χρειαζόταν ε, δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε έτσι ξαφνικά, είναι αδικαιολόγητο. Έχω την αίσθηση ότι έχει επιτευχθεί πολύ σημαντική πρόοδος μέχρι στιγμής. Βλέπω λοιπόν ότι το αν ανατρέξει κανείς ή αν μάλλον οπισθοχωρήσει, στην ουσία κάτι τέτοιο θα ζημίωνε την αξιοπιστία που έχει οικοδομηθεί μέχρι στιγμής και θα σήμαινε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό και από την αρχή θα δημιουργείται δηλαδή μια ένα η διαδικασία και αυτή είναι η άποψη της ΕΚΤ ότι πρέπει να, δούμε, να κοιτάμε μακροπρόθεσμα, να επιμείνουμε και δεδομένης της προόδου που έχει γίνει και της αξιοπιστίας που έχει επιτευχθεί μέσω αυτών των μέτρων οποιοδήποτε χαλάρωση ή δισταγμός θα ήταν αντι, αντιπαραγωγικός. Θα σήμαινε αυτόματα αύξηση των ε, επιτοκίων και εκ νέου έναρξη του αρνητικού κύκλου. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Θα τα πω τώρα αγγλικά για τα μήνυμα πιο σύντομα. Δεν λέω εγώ για να πάμε πίσω ή να οπισθοδρομήσουμε ή να μην κάνουμε, να μην έχουμε κάποιο είδου λιτότητα. Απλώς ισχυρίζομαι ότι η δόση είναι υπερβολική, το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό και το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά σύντομο. Από τη στιγμή που υπάρχει μείωση της οικονομικής ανάπτυξης, το νομικό κείμενο, το εξαπλό πακέτο, επιτρέπει ε, απαλότερη προσαρμογή. Ας το κάνουμε λοιπόν. Αντί να έχουμε δηλαδή περικοπή 130 δις ευρώ, μπορούμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα να το κάνουμε 80, να μειώσουμε 80-85, να ακολουθήσουμε δηλαδή τα νομικά κείμενα και να ε, καθυστερήσουμε το βήμα και την ισχύ όλων αυτών των μέτρων, γιατί όλοι οι υπολογισμοί των πολλαπλασίων είναι λάθος. Εφόσον ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τη συνταγή αυτή πια, Πολιτικά λοιπόν είναι πολύ λεπτό το θέμα. Περί αυτού λέω. Και δεν είπα να ξεχάσουμε την επιθαρχία και να οπισθοδρομήσουμε, να προσαρμοστούμε ώστε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Θα είμαι πολύ σύντομο στην απάντησή μου. Εκεί όπου υπάρχουν πολύ μεγάλα ελλείμματα προπολογισμού δεν υπήρχε ούτε τότε ανάπτυξη. Δεύτερη, πρώτη απάντηση και δεύτερη απάντηση και κάτι που με ρωτήσατε και πριν και δεν το απάντησα. Για τα κέρδη της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ τα μοιράζει τα, τα κέρδη τη. Αυτή είναι απόφαση των μελών. Δεν είναι απόφαση τη ΕΚΤ. Τα διανύμει στα μέλη της SCB και εκείνοι με απόλυτη ανεξαρτησία τα μοιράζουν στις κυβερνήσεις τους που με τη σειρά τους αποφασίζουν τι θα κάνουν αυτά τα κέρδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Ελίσσα έβγαλε πολύ ζωμή μέσα από αυτά τα πέντε λεπτά που είχε στη διάθεση η κυρία Σιλβί Γκουλάχ από το Άλτε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα για τη δημοκρατική νομιμότητα και την έννοια αυτή που είχε περιληφθεί στις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου του Ιουνίου. Ε, σημασία σε αυτό το θέμα είχε δοθεί, αλλά όχι αρκετή όπως αυτή που είχε δοθεί στο έγγραφο του κυρίου Ρομπόετ συμφωνείτε με τη δική μου μεγάλη απογοήτευση ως προς το θέμα αυτό, το οποίο δεν είναι καθόλου ίσονος σημασίας και δεν θα πρέπει να το διατρέχουμε εντάχει στο τέλος του εγγράφου. Γιατί συχνά τα επίσημα έγγραφα δίνουν την αίσθηση ότι καταληκτικά στην τελευταία παράγραφο κάνουν και μια αναφορά στο θέμα αυτό για τα μάτια του κόσμου. Από εκεί και πέρα, έχω την αίσθηση ότι αυτό που μας χρειάζεται είναι πολιτικές τις οποίες θα αποφασίζουμε από κοινού, βασιζόμενοι στη δημοκρατική διαδικασία και οι οποίες θα ισχύουν ε, για όλους. Βλέπω ότι σας σερβίρουν καφέ κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα να μην τον πάρετε, δεν είναι και πολύ καλός. Εν πάση περιπτώσει, Συνεχίζω λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο προτείνει το Συμβούλιο να αγωνιστούμε εναντίον αυτή της, της κατάστασης μου φαίνεται ότι αντίκειται ε, στην κοινοτική μέθοδο. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, κρίσιμη στιγμή είναι η ώρα που ε, έρχεται ο καφές. Ο κύριος Ντράγκη. Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι όλα τα βήματα είναι βήματα προς τα εμπρός και το Συμβούλιο του Ιουνίου ήταν ορόσημο για την επανεκκίνηση του ευρώ, για την παγίωση της ε, νομισματικής ένωσης. Από εκεί και πέρα συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Θα πρέπει η διαδικασία αυτή να συνοδεύεται από την δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία και βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστεί η εργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουλάχ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα άλλο τον κύριο Πρόεδρο. Μου αρκούν αυτά που είπε. Καλώς λέει η Πρόεδρος, ο Ντέρκ Γιανέπικ από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με τις ε, εκθέσεις του τύπου, οι νομικοί της Bundesbank είδαν ότι τα σχέδια για την Τραπεζική Ένωση στερούνται επαρκούς νομικής βάσης και εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη σαφήνειας ως προς τις εξουσίες του νέου υποπτικού μηχανισμού ε, και ε, επιφυλάξεις ως προς την Επιτροπή Συνδιαλλαγής, η οποία έχει ως σκοπό να διευκολύνει όλη αυτή τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και δίδεται ιδιαίτερη σημασία εσείς στις απόψεις της Bundesbank και αυτό σας καλώ να σχολιάσετε αυτά τα δημοσιεύματα. Ευχαριστώ. Απάντηση. Κοιτάξτε, οι δικηγόροι της Bundesbank είναι εξαιρετικά καλοί, αλλά έχουμε και εμείς νομικού συμβούλους, έχει και επιτροπή. Ε, και όλοι με τις διάφορες αποχρώσεις έννοιες τους και ειδικότητε και εξειδικεύσεις τους έχουν δώσει το πράσινο φως για το ε, πόσο ισχυρά είναι τα νομοθετικά θεμέλια αυτής της πρότασης. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει, ε, αν θέλετε, μια πιο παθητική στάση. Ε, εμείς εκφράζουμε γνωμοδοτήσεις επί της απόψης των άλλων είμαστε το υποκείμενο που δέχεται, όχι αυτό που στέλνει. Από την οικονομική σκοπιά όμως και από τη διαχειριστική σκοπιά αλλά και τη νομική εμείς θεωρούμε ότι όλη αυτή η άποψη έχει νομικά θεμέλια, είναι βασισμένη ε, σε επαρκή νομική βάση και θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και εγκαίρως να παρέχουμε αυτό τον εποπτικό μηχανισμό. Ευχαριστώ. Ο Φίλιπ Λάμπερτς για τους Πρασίνους τώρα. Ε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, καλώς ήλθατε και πάλι στις Βρυξέλλες. Δύο ερετήσεις. Πρώτον για το SSM το Κοινοβούλιο ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν έχει διαιρεθεί η αρμοδιότητα για την εποπτεία. Δηλαδή πάντα ένας παίκτη θα την έχει, δηλαδή εσείς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρωταρχικές αποστολές εποπτείας θα τις αναλάβουν οι εθνικές εποπτικές αρχές, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορεί να καλέσει ατομικά όποια τράπεζα επιθυμεί και θα το θεωρήσει σκόπιμο να κάνει κάτι τέτοιο. Σας ικανοποιεί αυτή η ρύθμιση από τη στιγμή που γνωρίζετε... Ε, ότι δεν θέλουμε διαίρεση της τραπεζικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί συμφωνούμε. Η Τραπεζική Ένωση δεν είναι ουσιαστικά δύο τραπεζικές ενώσεις. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Κατά δεύτερο λόγο, ο Μακάρνι και άλλοι έχουν τοποθετηθεί επ' αυτού. Δηλαδή η επιδίωξη της καταστολής του πληθωρισμού δεν θα πρέπει να είναι η μόνη αιμονή μιας κεντρικής τράπεζας. Ενδεχομένως θα πρέπει να επιδιώκει και στόχους ε, επίτευξης και βελτίωσης των δικτών μακροπρόθεσμης απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Ποια η άποψή σας επ' αυτού απάντηση. Ως προς το πρώτο συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Με το βήμα αυτό θέλουμε να έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα, μία τραπεζική ένωση. Εμείς θα εποπτεύουμε το σύνολο των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ε, θα εφαρμοστεί αυτή η εποπτεία θα είναι διαφορετικός αναλόγως με το μέγεθος του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Επομένως, η συμφωνία περιλαμβάνει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και έτσι μιλούμε για 100 με 300 τράπεζες που θα είναι υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ οι υπόλοιπε θα είναι 100 μέχρι, ε, μάλλον διορθών, 130 με 150 διορθών θα είναι υπό την άμεση, τραπεζική, ε, υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι υπόλοιπες ε, εμέσως. Τι θα συμβεί όμως σε γενικές γραμμές και αυτό επιβάλλει και η κοινή λογική η εποπτεία θα γίνεται όλο και πιο στενή όσο πιο κοντά φτάνουμε στο κέντρο, στο πυρήνα, όσο πιο μεγάλη είναι μια τράπεζα. Και αντιστρόφως, ο ρόλος της Εθνικής Εποπτικής Αρχής θα ε, είναι μεγαλύτερος όσο μικρότερη είναι η τράπεζα σε εθνικό επίπεδο. Ούτως ή άλλως όλες οι υποπτικές αρχές θα υπόκεινται στους κανονισμούς, στα πρότυπα και στο ενιαίο ε, εγχειρίδιο κανόνων, το οποίο είναι ε, και στόχος μας να το εφαρμόσουμε κατά γράμμα και όλα αυτά θα ρυθμίζονται από το κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει την εξουσία, την αρμοδιότητα που έχει να καλέσει ατομικά οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και θα έχει και την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα, την εξουσία να θέσει οποιοδήποτε ερώτημα, να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφόρηση, οποιοδήποτε στοιχείο. Και εγώ διάβασα δημοσιεύματα στον τύπο, τα οποία ανέφεραν ότι με αυτό το σύστημα θα καταλήξουμε σε ένα κατακαιρματισμένο τραπεζικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την άποψη δεν συμφωνώ. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας τώρα, ε, το θέμα είναι το εξής καταλαβαίνω τι εννοείται όταν αναφέρεται τον κυβερνήτη κύριο Κάρνι, Μακάρνι, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι αυτός μιλάει σε ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Η, η Κεντρική Τράπεζα αυτή έχει εντολή όχι μόνο να μεριμνά για τη σταθερότητα των τιμών, αλλά και για να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, να μεριμνά για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, βελτίωσης της οικονομικής ανάπτυξης και Η Κεντρική Τράπεζα στην οποία αναφέρεστε έχει περισσότερες εντολές ε, τις οποίες θα πρέπει να φέρει σε πέρας κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Λάμπερτς, πιστεύετε ότι θα υπάρξει κίνδυνος οι τράπεζες να προσπαθήσουν να ξεφύγουν από αυτόν τον κανόνα των 30 δις στον ισολογισμό τους. Απάντηση. Όχι. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι τράπεζες δεν ξεφεύγουν από το όριο αυτό. Δηλαδή η Εθνική Εποπτική Αρχή εποπτεύει το σύνολο του ισολογισμού των τραπεζών. Δεν θα αλλάξει αυτό τώρα. Δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει το σύστημα εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το σύνολο μιας τράπεζας θα την χάνει εποπτείας. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ η Μαρίσα Ματίας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ντράκη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας για να σας θα απευθύνω το ερώτημά μου. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω τα εξής ερωτήματα. Είναι γεγονός ότι κάθε φορά που κάνετε μία παρέμβαση, πάντοτε αναφέρεστε ε, στο ίδιο θέμα. Ωστόσο, λείπει η αλληλεγγύη. Λέτε καλά λόγια για την Τραπεζική Ένωση, αλλά δεν λέτε ότι αν αποτύχει αυτή η Τραπεζική Ένωση θα είναι πάλι ο σώζον αυτόν σωθήτο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντοτε μιλάτε για ε, το καλό σενάριο, εκεί όπου τα πράγματα λειτουργούν, αλλά δεν αναφέρετε τι θα γίνει όταν υπάρχει αποτυχία. Βλέπετε ότι τα σχέδια διάσωσης παρεκκλίνουν, φεύγουν, ε, εκτροχιάζονται και αυτό γίνεται ξανά και ξανά. τελικά δεν λύνεται το θέμα του χρέους. Μιλάτε για τις εξαγωγές και την αύξησή τους. Πράγματι, αυξήθηκαν κάπως οι εξαγωγές στις χώρες του Νότου, στην Πορτογαλία και στις άλλες χώρες που έχουν μπει σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό οφείλεται όμως και σε άλλους παράγοντες. Οφείλεται και στον στρατηγικό ρόλο που μπορεί ε, να έχουμε εμείς ως Πορτογαλία π.χ. με τη Βραζιλία, ε, με τις εμπορικές μας σχέσεις μπορεί να οφείλεται στην ε, ραχδαία αύξηση της ανεργίας. Με δεδομένο λοιπόν ότι το έλλειμμα και το χρέος θα συνεχίσει να εκτροχιάζεται και να είναι μεγέθη που εκτροχιάζονται αυτά συνεχώς στη χώρα μας μεταξύ άλλων χωρών, θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Ο κύριος Λάγεν παρακάλεσε η ομιλήτρια να μιλάει όχι πιο αργά αλλά πιο χαμηλόφωνα και η πρόεδρος σημειώνει ότι μάλλον φταίνε τα μικρόφωνα. Θα τα ξαναπώ από την αρχή και δεν θα μιλάω τόσο δυνατά. Αυτό που έλεγα και θα μιλήσω πιο δυνατά. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ κύριε Δράγκη, υπάρχουν δύο ερωτήματα που θέλω να μου απαντήσετε. Το ένα είναι πολύ προφανές. σε όλα τα σημαντικά θέματα, τα δύσκολα. Όχι, τι έγινε. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν έχουμε διερμηνία, μισό λεπτάκι. Μπορώ να τα πω και αγγλικά. Λοιπόν, τρίτη και τυχερή ελπίζω. Καταρχήν σας ευχαρίστησα που ήρθατε και το δεύτερο ε, θέλω να σας ε, ε, κάνω δύο ερωτήσεις για δύο παραδείγματα που δώσατε γιατί σε όλες τα δύσκολα θέματα που έρχεστε και μας παρουσιάζετε υπάρχει πάντα μία διάσταση όπου τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν τα καταφέρνουν και έχει να κάνει με την αλληλεγγύη. Και αν αυτό ισχύει σε ένα παράδειγμα που είναι η Τραπεζική Ένωση, γιατί ένα από τα πράγματα που δεν μας λέτε είναι όταν όλα αποτύχουν το γεγονός ότι όλοι πάλι θα χωριστούν, θα πει ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός αλληλεγγύης. Το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να μιλήσω είναι τα προγράμματα διάσωσης. Κύριε Ντράγκη, εσείς έρχεστε πάντοτε εδώ, έρχεστε πάντοτε εδώ και μας λέτε πως ήταν επιτυχή. Αλλά δεν ήταν επιτυχή. Οι βασικές μεταβλητές, το έλλειμμα και το χρέος είναι εκτός ελέγχου και συνεχίζουν να είναι εκτός ελέγχου. Ποια είναι η συνταγή σας, ότι δηλαδή κάθε φορά που οι μεταβλητές που είναι ο βασικός στόχος των ε, προγραμμάτων διάσωσης ε, βάζετε και άλλους στόχους εκτός ε, άσχετες, άσχετες παραμέτρους όπως οι εξαγωγές. Για παράδειγμα, γιατί στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κάπως οι εξαγωγές, αλλά το εμπορικό ισοζύγιο είχε να κάνει με την μείωση των εισαγωγών και όχι τόσο με την αύξηση των εξαγωγών. Ναι, σταματήσαμε το ρολόι με τα προβλήματα αυτά και εσείς μιλήσατε για 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Οπότε Μάριο πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος. Ναι, ευχαριστώ. Για το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, ε, ο εποπτικός μηχανισμός έχει όλες τις ε, εξουσίες για να είναι αποτελεσματικός. Η πρόκληση είναι λοιπόν η εφαρμογή του. Και γι' αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πως είναι ένα πρώτο μήνυμα για μια τραπεζική ένωση. Υπάρχουν δύο ακόμα βήματα. Το ένα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού ε, διάλυσης ή εξαγοράς τράπεζας και πάλι αυτό περιλαμβάνεται στα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στα συμπεράσματα και την επόμενη χρονιά η Κομισιόν θα υποβάλει σχετική πρόταση και το τρίτο σκέλος είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ε, ασφάλισης ε, καταθέσεων. Αυτό σημαίνει αμοιβεοποίηση του κινδύνου, κοινή μοιρασιά του κινδύνου. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και ο μηχανισμός εποπτείας είναι ένα από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στις τράπεζές μας, άσχετα από το πού βρίσκονται που είναι εγκατεστημένε. Δεύτερο σκέλο είναι περισσότερο δήλωση και όχι ερώτηση. Είπατε ότι το, το, το χρέος και το έλλειμμα είναι εκτός ελέγχου. Κατά με δεν είναι εκτός ελέγχου. Υπάρχουν ουσιαστικά προγράμματα. Είμαι βέβαιος ότι έχει υπάρξει πρόοδος με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρόεδρος, συγγνώμη, έχει τελειώσει ο χρόνος και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος ο Μάριο να επεκταθεί, να επανέλθετε. Σαμποτέρχο από την Ιευδίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ε, έγινε πολλή συζήτηση σε σχέση με τους διάφορους ρόλους της ΕΚΤ. Εσείς κάνατε κάποιες παρατηρήσεις στην εναρκτήρια ομιλία σας επίσης. Τώρα η ΕΚΤ πρέπει να αποδώσει και να λειτουργήσει ως υπεύθυνη αρχή για την νομισματική πολιτική καθώς και ως επόπτη των τραπεζών. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει καταμερισμός ε, καθηκόντων στο προσωπικό σας. Ε, ο πρόεδρος πώς θα τα καταφέρει. Το ερώτημά μου είναι πώς ε, έχετε σχεδιάσει πώς ο προσωπικός σας ρόλος ή το, η θέση στην οποία κατέχετε θα οργανωθεί στην νέα ΕΚΤ. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ελέγχει και τα δύο αυτά έργα. Πώς θα το οργανώσετε αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, αλλά δεν θα το ρυθμίσω εγώ αυτό. Θα υπάρξει μια τελείως ξεχωριστή αρχή, δηλαδή το εποπτικό συμβούλιο με διαφορετικό πρόεδρο και αντιπρόεδρο και ούτω καθεξής. Και αυτό θα λαμβάνει τις αποφάσεις του με πολύ ανεξάρτητο τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο και θέλουμε έτσι να μείνουν τα πράγματα διότι όπως έχω πει επανελειμμένως ο κεντρικός στόχος της ΕΚΤ είναι να διατηρεί την σταθερότητα των τιμών. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά για τα οποία μίλησα την πρώτη φορά που χρειάστηκε να μιλήσω δημόσια για αυτό το θέμα. Ό,τι και αν προκύψει είχα πει θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η νομισματική, η πολιτική και η εποπτεία θα είναι αυστηρά ε, διαχωρισμένες. Θέλετε να επανέλθετε με περώτηση, όχι. Ευχαριστώ, σα ευχαριστώ. Τώρα δεν έχω κανένα μία γεγραμμένο εδώ, οπότε εξ του ΕΛΚ η Μαριάν Τάισεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω εισηγήτρια για τον μηχανισμό εποπτείας θα μου επιτρέψετε να σα κάνω ορισμένε ερωτήσει. Όπω και εσεί, αλλά και διάλφοι φαίνεται πώ σημειώνεται πάλι ένα πρόβλημα με την διερμηνία. Ίσως όμω δεν είναι τα ακουστικά. Μου φαίνεται ότι κάνω, κάναμε λάθος με τα κουμπιά, λέει η πρόεδρος. Αρχίστε πάλι αν θέλετε, σας παρακαλώ, αρχίστε πάλι. Να, να μιλήσω αγγλικά καλύτερα, λέει η κυρία Τάισιν. Ως, ε, στα αγγλικά λοιπόν. Oh. <laughs> Okay. Yeah. Mag ik nog eens opnieuw proberen? Να δοκιμάσω πάλι. Καλά λοιπόν, τότε θα αρχίσω πάλι στα φλαμανδικά. Είμαι εισηγήτρια λοιπόν για το θέμα του μηχανισμού εποπτείας και θα ήθελα να κάνω ορισμένε ερωτήσεις Χαιρόμαστε πρώτα που υπάρχει ενιαίος μηχανισμός εποπτείας. Ένα από τα θέματα, ωστόσο, που τίθεται είναι ότι το εποπτικό αυτό όργανο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να εκδώσει κατευθυντήρες γραμμές για τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Αλλά αυτές δεν μπορούν παρά να είναι γενικές κατευθυντήρες γραμμές. Εξάλλου, είναι δυνατόν να εκδοθούν και ατομικές καθευτηρίες γραμμές για συγκεκριμένες εθνικές αρχές όταν δεν λειτουργούν τόσο καλά. Αυτό θεωρείται ότι, πρόκειται, ότι είναι κενό ή θεωρείται ότι έχετε επαρκείς δυνατότητες από ό,τι σας ε, δίδουν οι σχετικές διατάξεις. Επίσης, αναβλήθηκε η θέση σε ισχύ. Εμείς είχαμε θεωρήσει ότι θα άρχιζε από 1η Πρώτου 2014, να τώρα αρχίζει από 1η Μαρτίου 2014. Και φαίνεται τώρα επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ακόμα έτοιμη για την εφαρμογή του. Εάν διαπιστώσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν είναι έτοιμη ακόμη, μπορεί να αναβάλει την θέση ισχύ του μηχανισμού εποπτείας και πέρα από τον Μάρτιο του 2014. Η... Αυτή είναι η κυρίως η ερώτησή μου. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και την πολιτική σας ομάδα για την δουλειά που κάνατε και που έθεσε και τα θεμέλια για τις αποφάσεις. Θέτεται εδώ δύο ερωτήματα. Αφενός οδηγίες, γενικές οδηγίες ε, ως αντιπαρατίθεται στις ειδικές ή ατομικές οδηγίες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να εκδώσει γενικές οδηγίες προς τους εθνικούς επόπτες. Αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο για την έκδοση ειδικών οδηγιών, ατομικών οδηγιών. Δεν νομίζουμε. Είναι γεγονό ότι θα είναι γενικέ οδηγίε, αλλά μέχρι ενό σημείου. Δηλαδή, μπορούμε να εκδώσουμε οδηγίε για, ε, για κατηγορίες, ή ομάδες τραπεζών. Και όταν μιλούμε για οδηγίες, είναι δύσκολο να εκδοθεί μια οδηγία που να έχει κάπως γενική εφαρμογή, αλλά να εφαρμόζεται μόνο σε, μια συγκεκριμένη ή σε λίγες συγκεκριμένες τράπεζες. Μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με τις τράπεζες και με διαφορετικό τρόπο και όχι με την έκδοση οδηγιών. Αυτό λοιπόν δεν είναι σημαντικό το θέμα. Το άλλο είναι η θέση σε ισχύ, η πραγματική δηλαδή έναρξη λειτουργίας του εποπτικού μηχανισμού και του timing. Η ιδέα που έχουμε εδώ είναι ότι είναι σημαντικό να γίνει σύντομα, αλλά πιο σημαντικό ακόμη είναι να γίνει σωστά. Είναι αλήθεια ότι χρειαστήκαμε ένα χρόνο μετά από την θέση σε ισχύ του κανονισμού του Συμβουλίου Νομίζουμε λοιπόν ή υπολογίζουμε αν θέλετε καλύτερα ότι θα πρέπει να είναι τον Μάρτιο του 2014 εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των τριμερών διαλόγων καθώς επίσης και τεθεί ισχύ ο κανονισμός του Συμβουλίου. Θα μπορέσουμε τότε να αρχίσουμε τον Μάρτιο. Όμως προχωρούμε σε ε, εδάφη ή σε ύδατα όπου δεν ε, είναι άγνωστα. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια ευκαμψία για την περίπτωση όπου υπάρξουν απρόβλεπτα εμπόδια ή άλλα κολλήματα. Ας μην δυσμονούμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν και οι εθνικοί επόπτες. Για παράδειγμα, στατιστικές, αλλαγή εθνικών νομοθεσιών, χορήγηση, δηλαδή αίτηση και χωρί εκ μέρους τους ε, πολλών δεδομένων. Ε, γι' αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται κάποια, κάποιος χρόνος. Ευχαριστώ. Θέλετε να λάβετε ξανά το λόγο, Μαριάν. Ίσως μπορώ να επανέλθω με άλλη ερώτηση. Τότε σας μένει μόνο 45 δευτερόλεπτα. Ίσως να μην μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Δράγκη. Τα χρειάζεστε πριν από την θέση ισχύ του μηχανισμού. Χρειάζεται μόνο μια resolution authority, ε, δηλαδή ε, αρχή για τις ε, διαλύσεις των τραπεζών ή χρειάζεται και ταμείο. Αυτό έχει σχέση και με τα όσα είπα για το χρονοδιάγραμμα, το timing. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει και κάθε ενδιαφέρον να ε, ιδρυθεί σύντομα και να λειτουργήσει ο εποπτικός μηχανισμός. Για τον ενιαίο μηχανισμό διαλύσεων και εξαγορών, η ιδέα είναι ότι τα δύο αυτά πράγματα θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν πλήρως μαζί, ταυτόχρονα. Και επειδή ο ενιαίος μηχανισμός διαλύσεων είναι πολύ σημαντικός γιατί μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε πτωχεύσεις τραπεζών που ενδέχεται να, να συμβούν με τρόπο που, δεν, που μας επιτρέπει να μην χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων και ταυτόχρονα ε, δεν καταστρέφει μεγάλα τμήματα του συστήματος πληρωμών, πράγματα τα οποία είδαμε να συμβαίνουν στη διάρκεια της ε, δημοσιονομικής κρίσης. Είδαμε δηλαδή ε, πτωχεύσεις τραπεζών, οι οποίες, καταρρεύσεις τραπεζών, οι οποίες είχαν και τις δύο αυτές συνέπειες, δηλαδή και διάσωση με χρήματα φορολογουμένων και ε, καταστροφή τμήματων του συστήματος πληρωμών. Αυτό λοιπόν είναι, μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε και ενδεχόμενες των τραπεζών, κυρίω αυτών που έχουν έδρα σε, σε πολλές χώρες και που τώρα ε, βρίσκονται υπό διαφορετικά ε, νομικά καθεστώτα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πρώτα το νομοθετικό τμήμα και μετά θα δούμε ενδεχομένω και το Ταμείο και, την Ανεξάρτητη Αρχή. Βέβαια το ιδεώδε θα ήταν όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν ταυτόχρονα. Ο Βέρνερ Λάνγκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εγώ παρακολουθώ πάντοτε με πολύ θετικό πνεύμα και αξιολογώ με θετικό πνεύμα την εργασία σας. Τώρα όμως όπως εξηγήσατε, αναλαμβάνετε την ευθύνη εποπτείας όλων των τραπεζών. Εγώ βρίσκω να υπάρχουν πολλά προβλήματα εδώ. Πρώτη μου ερώτηση, ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες αναθεωρήσεις στα ε, κείμενα των συνθήκων. Το άρθρο 127 παράγραφος 3 του καταστατικού της ε, τράπεζας προβλέπει τις λειτουργίες αυτές και προβλέπει ε, και στο άρθρο 25 και ε, την διαδικασία. Άρα δεν υπάρχει λόγος αναθεώρησης. Ο κύριος Σάλμπα επίσης ρώτησε, και εδώ είναι η δεύτερη μου ερώτηση, το πρόγραμμα χρημάτων που ανέχεται σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα χρήματα που διατέθηκαν δηλαδή, είχαν διαφορετική, διαφορετικά αποτελέσματα. Οι νότιο-ευρωπαϊκές τράπεζες δεν έδωσαν χρηματοδοτήσεις και προτίμησαν να αγοράσουν ομόλογα. Και αυξήθηκε η χρέωση των τραπεζών ε, Ισπανίας, Ελλάδας, Ιταλίας κατά 99%. Επίσης, τρίτο ερώτημα. Πώς θα γίνει ο χωρισμός όταν τέσσερις από τους έξι ε, Διευθυντέ τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μέλη και σε αυτά τα όργανα. Πρόεδρος Δράγκη, μια διόρθωση για το τελευταίο αυτό δεν είναι αληθές. Προβλέπεται το Supervisory Board να είναι από τους, να, συνδίθεται από τέσσερα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά σύν του Επόπτε των ε, χωρών μελών, συν ενδεχομένως και τι νέε χώρε οι οποίες θα μπουν στην επιπτικό μηχανισμό, εκτός, ευρώ, εκτός δηλαδή ζώνη ευρώ. Δεν πρόκειται λοιπόν να είναι τα ίδια πρόσωπα. Για το δεύτερο θέμα που θίξατε, για τα χρήματα που διατέθηκαν για να αγοραστούν κρατικά ομόλογα. Αυτό είναι εν μέρη ορθό. Η χρήση που έκαναν οι τράπεζες της ρευστότητας που έλαβαν από τον LTRO ήταν να ξεπληρώσουν τα, τα δικά τους ομόλογα. Μην λησμονούμε ότι 230 εκατομμύρια κρατικών ομολόγων επρόκειτο να οριμάσουν στο πρώτο τρίμηνο του φετινού χρόνου. Έτσι λοιπόν απεθεύθη μια μεγάλη κρίση και βεβαίως αγόρασαν μετά και κρατικά ομόλογα. Και το θέμα είναι, νομίζω ότι το συζητήσαμε σε άλλη ευκαιρία αυτό, το ερώτημα είναι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποτρέψει τι τράπεζε αυτέ από το να αγοράσουν κρατικά ομόλογα και να τι να, να τις αναγκάσει να, να την οικονομία. Η απάντηση που δίνω εγώ πάντοτε σε αυτήν την ερώτηση είναι ορισμένοι λένε πρέπει να, δώσουμε, να αναγκαζέσουμε τις τράπεζες να δώσουν λεφτά στην οικονομία και οι άλλοι που λένε να φροντίσουμε ώστε οι τράπεζες να μην αγοράσουν κρατικά ομόλογα ζητούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να κάνει κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Να πει δηλαδή στις εθνικές τράπεζες τι θα κάνουν με τα χρήματά τους. Τώρα, για να τις προτρέψουμε να δανειοδοτήσουν την οικονομία, νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά πράγματα. Για παράδειγμα, με την ανάπτυξη των ασφαλιών, με, του collateral. Και επίσης βάλαμε τις τράπεζες σε μια κατάσταση όπου όσο περισσότερο δανείζουν, τόσο περισσότερο collateral έχουν για να χρηματοδοτήσουν με την βοήθεια της Κεντρικής Τράπεζας. Εάν σκεφτείτε όμως ποια είναι η περιπλοκή που θα ε, συνεπάγεται κάθε πρόγραμμα το οποίο θα λέει στις τράπεζες τι να κάνουν σε μια ε, ζώνη ευρώ με 17 χώρες μέλη. Δηλαδή θα πούμε στις τράπεζες θα σας, δώσουμε, θα σας δανείσουμε χρήματα μόνο αν δανείσετε και παραπέρα στην οικονομία. Τότε αυτό πρέπει να εξετάσουμε, να το διερευνήσουμε αν είναι αληθές. Είπαμε 600 τράπεζες ή 150 οι οποίες επανήλθαν τον Μάρτιο για να δανειστούν από τον LTRO. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές περιπλοκότητες αυτών των προγραμμάτων που είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Τώρα για το πρώτο σας θέμα για τα νομικά θεμέλια. Νομίζω ότι απάντησα προηγουμένω. Δεν είμαι νομομαθή, ή δικηγόρος, πρέπει να εμπιστευτώ άλλου νομομαθεί που μου λένε ότι είναι στέρεα τα νομικά θεμέλια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να δούμε οι ίδιοι πώς ερμηνεύουν το άρθρο 127 παράγραφος 6. Εγώ δεν θα προβώ σε άλλα σχόλια, παρά μόνο ότι στο προκείμενο βασίζομαι στην κρίση άλλων. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις ανησυχίες του Πέρναν Λάγκεν για το πώς θα διοχετευτεί το χρήμα στην πραγματική οικονομία. Οι κεντρικές τράπεζες ε, καθοδηγούσαν, αλλά τελικά απέσυραν τη στήριξή τους και εμέσως κάθε τράπεζα ε, ε μπορούσε να προσφέρει εγγύησεις. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Αντολίν Σάντσεφ Περεσέδο για τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την ε, στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας φέτος. Μου έλειπε στο παρελθόν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπέζα παλαιότερα δεν συνέβαλε σε αυτή την δημοσιονομική ε, θεσμική προοπτική και τώρα το κάνει περισσότερο. Πώς μπορεί να συμβάλλει στους βασικούς μας στόχους. Και οι βασικοί μας στόχοι γνωρίζετε ότι είναι η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σήμερα μάλιστα που συρρυκνώνονται οι οικονομίες μας διότι συρρυκνώνονται και οι γραμμές πίστοσης. Επομένως, ως προς τις χώρες που μπορούν να τύχουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα ομόλογα τους δηλαδή. Θα μπορούν να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρώτον. Και δεύτερον με την άμεση ανακεφαλαιοποίηση. Φαίνεται ότι είναι απαραίτητο. Ε, τα προγράμματα που έχουν άμεση στήριξη ε, πώς μπορεί εκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει καλύτερη εποπτεία. όπω uh, Όπως είπα και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, λέει ο κ. Ντράγκη, πράγματι η φετινή χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Εάν ανατρέξουμε στο παρελθόν και δούμε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όλη αυτή τη χρονιά, τότε σίγουρα θα συμπεράνουμε ότι πράγματι αναλάβαμε δράση με πολύ ενεργητικό ε, ρυθμό. Χαμηλώσαμε τα επιτόκια τρεις φορές. Κάναμε δύο φορές τα LTRO. Επιβάλαμε το collateral. Συζητήσαμε τον λόγο για τις ελάχιστες κεφαλαϊκές απαιτήσεις ε, των τραπεζών, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια βεβαίως. Αναλάβαμε ένα σωρό δράσεις δηλαδή μέχρι την ανακοίνωση του Ιουλίου για το OMT. Άρα καταφέραμε να πετύχουμε σταθερότητα τιμών σε μεσοπρόθεσμη βάση, εάν εξετάσει κανείς και την πορεία και τη διακύμαση του πληθωρισμού και κατά πόσο ε, είναι σταθερές οι προσδοκίες για το μακροπρόθεσμο πληθωρισμό. Εν πάση περιπτώσει όμως, όλη αυτή η ρευστότητα πρέπει να φτάσει στην πραγματική οικονομία και για να γίνει αυτό χρειάζεται χρόνος. Η τρέχουσα κατάσταση ε, δείχνει ξεκάθαρα πόσο σοβαρή ήταν η κρίση χρηματοδότησης η οποία ξέσπασε ε, και έφτασε σε μεγάλη κλίμακα την περασμένη χρονιά. Τα δύο LTRO, οι δύο αυτές επιχειρήσεις, αν θέλετε, λειτουργίες μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, ε, κατέφεραν να αποφύγουμε ακόμα ακόμα, μια ακόμα πιο σοβαρή κατάσταση. Δεν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να σπρώξει τις κυβερνήσεις να υποβάλουν αίτημα για τέτοιου είδους βοήθεια. Οι κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια ξέρουν πολύ καλύτερα τα ίδια τι να κάνουν και πότε να το κάνουν όπου αυτό και όποτε αυτό χρειάζεται. Ως προς την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η απόφαση είναι η εξή. Μπορεί ο μηχανισμός σταθερότητας να ανακεφαλοποιήσει άμεσα τις τράπεζες μόνο και εάν θα υπόκειται στην εποπτεία λειτουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Σε επίπεδο Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ έχει τεθεί το θέμα των legacy assets και θα πρέπει να τα ορίσω αυτά τα στοιχεία ενεργητικού ε, που είναι κληρονομιά αν θέλετε και δεν είναι αυτό καθήκον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να τα προσδιορίσει ε, σε ποιο εύρος εκτείνονται. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος κυρία Μπόουλς. Καλώς Προχωρούμε με την Κορίν Βόρμαν Κόλ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντράγκη. Θα ήθελα να σας απευθύνω ένα ερώτημα ως προς την πρόοδο που έχουμε επιτύχει ε, για την, ε, ώστε η ΟΝΕ να μπει πάλι σε σωστή τροχιά. Έχετε νέα όπλα, μπαζούκα θα τα έλεγα, ε, και είναι αρκετά ικανά. Αυτό πάντοτε το λέγατε, αλλά πάντοτε λέγατε επίσης ότι θα πρέπει και οι πολιτικοί να δράσουν. Εξήρατε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου, υπογραμμίσατε την ανάγκη επίτευξης περαιτέρω προόδου για την ε, περαιτέρω ενοποίηση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής και ένωσης. Παρ' όλα αυτά, οι μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά που αναφέρατε στην εισαγωγή σας ε, δεν αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ερωτώ λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπό τις ε, συνθήκες, εάν οι συνθήκες είναι οι σωστές, είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει αυτό το νέο εργαλείο, το ONT, Είπατε ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν το ζητήσουν τα κράτη-μέλη, αλλά δεν θα το συνδέσετε με ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης ή εν μια σύμβαση, μια δέσμευση του κράτους ότι θα αναλάβει μεταρρυθμίσεις. Σχετίζονται αυτά με την ολοκλήρωση της ε, Οικονομικισματικής και Νομισματικής Ένωσης. Πιστεύετε ότι η πρόοδος στο Συμβούλιο είναι επαρκής και ενθαρρυντική με αυτή την, προς αυτή την κατεύθυνση μιας πραγματικής ονέ. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ε, κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές πρέπει να πω ότι όποια πρόοδος και αν σημειώνεται προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής οικονομικής και νοσηματικής ένωσης, αυτή θα σχετίζεται άρρηκτα με την ανάληψη δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικές ή και διαρθρωτικές, όπου δει. Όλα αυτά είναι σε σύνδεση με τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και μάλιστα αυτές οι συμβάσεις, οι δεσμεύσεις σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις με έμεσο τρόπο έστω, αλλά συνδέονται όλα αυτά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο η αγορά προϊόντων και η αγορά εργασίας είναι συμβατή με ε, την ύπαρξη μιας ε, οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία ε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ό,τι και να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ω προ το ΕΝΤ, ε, για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητε προποθέσει. Είναι μια απαραίτητη προπόθεση, υπάρχει αιρεσιμότητα η οποία είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκή, γιατί χρειαζόμαστε και ανεξάρτητη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ESM θα καθορίσει την αιρεσιμότητα. Θα πρέπει οι χώρες να υποβάλουν ε, αίτημα και θα πρέπει να παρέμβει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εάν τελικά συνεχίσει να είναι παρόν. Θα με εξέπλητε λοιπόν, εάν τελικά καθιερωθεί αυτό το πλαίσιο με τις ε, δεσμεύσεις και συμβάσεις για τη μεταρρύθμιση, για τις μεταρρυθμίσεις, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι πάντοτε θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα υπόλοιπα, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, η Κορίν θέλει ε, να κάνει υπερώτηση. Ναι, αυτό σχετίζεται με πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, αλλά γενικώ μιλάω για την, προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής νομισματικής ένωσης η πρόοδος θα πρέπει να είναι φιλόδοξη για να φτάσουμε εκεί. Είναι φιλόδοξη κατά την άποψή σας. Απάντηση. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά ήταν αρκετά καλή. Ας ανατρέξουμε στο παρελθόν, ας αναρωτηθούμε πώς ήταν η κατάσταση ακριβώς τον περασμένο Φεβρουάριο. Έκτοτε έχουν γίνει σημαντικά βήματα και από διάφορους θεσμικού φορείς και πρώτα απ' όλα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επομένω, εάν συγκρίνουμε ε, το 2012 με το 2011 π.χ. βλέπουμε ότι το 2012 είναι πράγματι μια χρονιά σημαντικής προόδου σε όλα τα μέτωπα προς μια ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, προς μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται ε, στα κράτη-μέλη και από πλευράς δημοσιονομικής και από πλευράς διαρθρωτικής, ενώ έχει γίνει και μεγάλη προόδος για τη σταθεροποίηση των ε, χρηματαγορών και χρηματοπιστωτικών αγορών γενικότερα. Ευχαριστώ. Η Αρλίν Μαρκάρθη από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Να επανέλθω στο ερώτημα του Φιλίπ Λαμπέρτς, γιατί επανειλημμένος στον τύπο έχετε πει ότι είστε παθητικός δράστης σε όλη αυτή τη συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλαδή, και ότι θα διατηρήσετε τη συνοχή ε, της ΕΚΤ με αυτό τον ενιαίο αποπτικό ρόλο που έχω ε, που έχετε. Αυτό το οποίο με έχει μπερδέψει είναι το γεγονός ότι ξεκινήσαμε με 6.000 τράπεζες και τώρα θα εποπτεύσετε 150. Άρα 6.000 με 150 τις υπόλοιπες θα τις εποπτεύετε από κοινού με τους εθνικούς μηχανισμούς εποπτείας. Ε, πώς θα το κάνετε αυτό. Ε, θα επιμείνετε στην εφαρμογή του ενιαίου βιβλίου κανόνων εποπτείας. Και αυτό πώς θα γίνει με τις διαφορετικές εθνικές εποπτικές αρχές το Συμβούλιο απέρριψε την ιδέα της κοινή ανάληψης χρέους. Δεν πρόκειται να μοιραστεί το βάρος σε διαφόρους και διαφορετικούς όμους. Ε, πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Θα χρηματοδοτηθούν θα το χρηματοδοτήσουν μόνο οι τράπεζες, ο φορολογούμενος ε, θα ε, πληρώσει και άλλη μια φορά. Ε, όταν κάποια τράπεζα θα πρέπει να διαλυθεί να εξαγοραστεί. Ορισμένοι πιστεύουν ότι θα πρέπει η τράπεζα να μπει σε ένα εθνικό σύστημα ε, διάλυσης ή εξαγοράς ως προϋπόθεση για, να, ε, για την εποπτεία της. Έχω κάπως μπερδευτεί, έχω λίγες γνώσεις για το θέμα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν καθόλου γνώσεις για το θέμα αυτό και τελούμε ε, σε σύγχυση και θα ήθελα να τα διευκρινίσω όλα αυτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Απάντηση. Κοιτάξτε, όταν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένας παθητικός ε, δράστης, εννοώ ότι είναι από την πλευρά αυτού που υποδέχεται το προϊόν της νομοθετικής διαδικασίας, την οποία καθορίζετε εσείς από κοινού με το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης που έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, πράγματι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποδέχεται τις νομοθετικές εντολές που αποφασίζετε εσείς. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της εφαρμογής και της υλοποίησης, αλλάζει τελείως το πράγμα τότε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι συνθήκες ε, για να λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός. Προχωρούμε λοιπόν μαζί. Μαζί αποκινούμε τις εθνικές εποπτικές αρχές. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα θα απαρτίζεται καταρχάς και πρώτα απ' όλα από τους εθνικούς επόπτες. Και όταν μιλώ για τις 150 τράπεζες, θέλω να σας πω το εξής. Νομίζει κάποιος κόσμος ότι θα μοιράσουμε την τραπεζική αγορά σε δύο κομμάτια και θα πούμε ότι το ένα κομμάτι το εποπτεύουμε εμείς στην ΕΚΤ και το υπόλοιπο το εποπτεύουν μόνο οι εθνικές αρχές. Δεν ισχύει αυτό. Είναι λάθος. Συνεργαζόμαστε. Δουλεύουμε μαζί. Ε, ο εθνικός μηχανισμός ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας είναι ένας μηχανισμός που θα ε, εφαρμόζουν και οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν έχουν ευθύνες για την νομισματική πολιτική. 150 τράπεζες θα τη χάνουν εποπτείας από το κέντρο και στις υπόλοιπες τράπεζες η εποπτεία από το κέντρο θα είναι λιγότερο κυρίαρχη και περισσότερο κυρίαρχη για αυτές θα είναι η εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών πάντοτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να εκδώσει οδηγίες για ομάδες ε, τραπεζών, αλλά ε, θα έχει και πάντοτε την αρμοδιότητα να καλέσει ε, συγκεκριμένη τράπεζα προκειμένου να υποβάλει περαιτέρω στοιχεία, πληροφορίες και το καθεξής. Άρα σε αυτές τις 150 τράπεζες ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσθεθεί συν άλλη μία οποιαδήποτε, εάν αυτό χρειάζεται. Και είναι ένα σύστημα το οποίο είναι εν τη γενέση του και το οποίο θα διαμορφώνεται στο βαθμό που θα εφαρμόζεται. Θα είμαι σε θέση να εξηγήσω περισσότερα όσο περισσότερο το εφαρμόσουμε και το τελειοποιούμε. Έρχομαι τώρα στο θέμα του Ταμείου ε, για την ε, ε, διάλυση εξαγορά των τραπεζών. 90 με 95% είναι νομικές αλλαγές και 5 με 10% είναι οι αλλαγές ως προς τα χρήματα. Πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο μηχανισμό για τη διάλυση ή εξαγορά τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να το ξεκαθαρίσω αυτό, να το εξηγήσω καλύτερα. Όταν κλείνει π.χ. μια τράπεζα, ε, η απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί είναι αν θα αναλάβουν μέρος του κόστους οι πιστωτές ή όχι. Ε, αν θα ε, σβήσουν εντός εισαγωγικών οι μέτοχοι ή όχι. Αυτός ο κατάλογος των πιστωτών αυτή τη στιγμή διαφέρει ε, ανά χώρα, από τη μία χώρα στην άλλη. Το να έχουμε έναν ενιαίο μηχανισμό για τη διάλυση ή εξαγορά των ε, τραπεζών σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε ή έχουμε συμφωνήσει ε, τι θα πρέπει να γίνει όταν κλείνει μια τράπεζα. Ποιοι είναι οι πιστωτές που θα συμμετάσχουν και τι θα γίνει με τους μετόχους και ποιο μερίδιο ευθύνης θα αναλαμβάνουν. Στη συνέχεια, χρειαζόμαστε ένα ταμείο για να τα διαχειριστεί αυτά. Δεν είναι ένα ταμείο διάσωσης της τράπεζας και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Εξού και το μέγεθος του ταμείου αυτού δεν θα είναι κατά ανάγκη τεράστιο θα είναι αυτό το οποίο ε, θα είναι απαραίτητο για να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις αυτές για τη διάλυση εξαγορά των τραπεζών. Π.χ. να κλείσουν κάποια υποκαταστήματα ή να χρηματοδοτηθεί η ε, μεταφορά της δραστηριότητας σε μια άλλη επικουρική, ε, η θηγατρική τράπεζα. Ε, συγγνώμη, έχω υπερβάλει κάπως γιατί παρασύρθηκα και πήρα περισσότερο χρόνο από ό,τι, έπρεπε. Η Πρόεδρος, ήταν και σημαντικά τα ερωτήματα. Να σας ρωτήσω το εξής. Δεν εποπτεύεται άμεσα κάποιες τράπεζες για τις οποίες η Εθνική Εποπτική Αρχή λέει όχι δεν θα μπουν στο καθεστώς διάλυσης ή εξαγοράς άρα θα πληρώσει ο φορολογούμενος. Εκεί τι θα κάνετε ως ΕΚΤ. Απάντηση. Καλό ερώτημα. Δεν έχουμε ακόμα απάντηση. Πρέπει να τη βρω την απάντηση. Δεν έχουμε προβλέψει κάτι για αυτή την περίπτωση. Έχω την αίσθηση όμως ότι η δήλωση του κεντρικού επόπτη, η οποία θα λέει ότι η χή τράπεζα πρέπει να κλείσει ή να εξαγοραστεί ή να διαλυθεί, εν πάση πτώση, είναι μια πολύ ισχυρή δήλωση και δεν αφήνει μεγάλο περιθώριο δράση στις εθνικές εποπτικές αρχές όποτε αυτή γίνει ως δήλωση. Ε, φανταστείτε το, την, τις επιπτώσεις όταν ε, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο πει ότι αυτή η τράπεζα ε, θα πρέπει να αλλάξει μορφή και τελικά οι εθνικές αποπτικές αρχές δεν κάνουν τίποτα. Τι νομίζω ότι θα κάνουν οι καταθέτες, θα αποσύρουν τις καταθέσεις τους οι αποταμιευτές. Άρα δεν νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα έχει ιδιαίτερο περιθώριο διαφοροποίησης η Εθνική Εποπτική Αρχή. Αλλά έχετε δίκιο, είναι καλύτερο να το έχουμε προβλέψει αυτό νομοθετικά και αυτή την περίπτωση εξ αρχής. Η Πρόεδρος, καλώς για το ΕΛΚ να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή για τις ε, προτάσεις αυτές. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις. Εσείς εξετά... παρουσιάσατε το πρόγραμμα της Κεντρικής Τράπεζας το Σεπτέμβριο και το Αμερικανικό ΦΕΔ προβλέπει 40 δισεκατομμύρια δολάρια τον ε, μήνα για επαναγορές και ανάλογα η Ιαπωνική τράπεζα. Αυτά έχουν κάποιες επιπτώσεις και βραχυπρόθεσμα και ηρεμούν τις αγορές. Θα ήθελα να μάθω από εσάς, αν κοιτάξετε και λίγο παραπέρα, τι κίνδυνο βλέπετε τονίσατε στην εισαγωγική σας ομιλία την ανάγκη να αποφευθούν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Βέβαια, μακροπρόθεσμα θα είναι, και γι' αυτό είστε αρμόδιος εσείς, πιο περίπλοκα τα πράγματα. και αν μπορείτε να πείτε και λίγα σχετικά με τον κίνδυνο κατακαιρματισμού ή και διάσπασης. Από το γεγονός ότι τώρα σχεδιάζουμε τον εποπτικό μηχανισμό στην βάση της ζώνης ευρώ των 17, αλλά κυρίως με ενδιαφέρον οι μακροοικονομικές συνέπειες. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω παρά μόνο για τη δική μου αρμοδιότητα αυτή, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εμείς ε, ε, κάναμε τους δύο, τις δύο φάσεις του μηχανισμού LTRO για την βελτίωση της ε, ρευστότητας. Κυρίως όμως η μείωση της έντασης προκλήθηκε από μια ανακοίνωση. Διακόπτη ο κ. Χέκμαρ. Ναι, αλλά τονίσατε ότι ήσασταν διατεθειμένο να αναλάβετε τις δράσει αυτές. Ναι, όσον αφορά τις δύο πρώτες αυτές επιχειρήσεις, είναι ότι δημιουργήθηκε μια βάση ε, χρήματο, αλλά δεν πήγε στο μη τρία. Για τον πληθωρισμό χρειάζονται τρία πράγματα. Να μην υπάρχει περιθώριο στην spare capacity και η ρευστότητα να περάσει στο μη τρία, δηλαδή σε πραγματικό χρήμα το οποίο να μπορεί να δαπανηθεί από τον κόσμο, διότι δανείζεται στον κόσμο, στους ανθρώπους. Δεν τα είδαμε αυτά, δυστυχώς. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και ταυτόχρονα, δυστυχώς κατά κάποιο τρόπο, διότι δεν κατέληξαν στους καταναλωτές τα χρήματα αυτά. Και ούτε, ούτε είδαμε και έλλειψη ε, και πάστη περιθωρίου ικανότητας δηλαδή είδατε ότι από 2,7% ο πληθωρισμό κατέβηκε στο 2,2%. Και μακροπρόθεσμα οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό φαίνεται να είναι σταθερές. Το επόμενο ερώτημα είναι τι θα γίνει αν πρόκειται να δούμε να συμβαίνει κάτι. Έχουμε πολλά εργαλεία που μπορούμε, που μας επιτρέπουν να μειώσουμε τη ρευστότητα που έχουμε δημιουργήσει πριν να μπει στο σύστημα και τέλη του έτους, αρχές του επόμενου έτους, θα δούμε ορισμένες τράπεζες να ε, ξεπληρώνουν τον LTRO, να επιστρέφουν δηλαδή τα χρήματα και έτσι να μειωθεί ο ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντιδράσαμε λοιπόν τον Ιούνιο, τέλη Ιουλίου, κατά του κατακαιρματισμού της ζώνης ευρώ, ευρώ που θα δημιουργούσε, θα προκαλούσε κάποια καταστροφικά σενάρια. Και σε κάποιο βαθμό από τότε είδαμε σαφή βελτίωση σε όλα τα μέτωπα στις οικονομικές αγορές. Τώρα, η έγκριση του επαπτικού μηχανισμού θα μειώσει ακόμα περισσότερο τον κατακαιρματισμό της ζώνης ευρώ. Η εντύπωση λοιπόν που έχει κανείς, τουλάχιστον για το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους, είναι μια σταδιακής βελτιώσεως των οικονομικών συνθήκων. Και για αυτό, αυτός είναι και ένας από τους λόγους για, τον για τους οποίους προβλέπουμε αρχή ανάκαμψης για το δεύτερο εξάμεινο του ε, επόμενου χρόνου. Η κυρία Ποδηματά. Σας ευχαριστώ Σάρων και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη διευκρίνηση σχετικά με το εάν τράπεζες που δεν ε, παρουσιάζουν συστημικό κίνδυνο και θα μείνουν σε εθνική εποπτεία θα επωφεληθούν ή όχι από την άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον ESM. Και δεύτερο, στα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου και παρά τις σημαντικές αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ που υποστήριξαν οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων για την ε, Τραπεζική Ένωση και για τον SSM ως πρώτο βήμα αυτού, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική ενοποίηση οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξες. Γι' αυτό ρωτώ, νομίζετε ότι η Τραπεζική Ένωση μπορεί να είναι πλήρως ενεργή, πλήρως λειτουργική, χωρίς μηχανισμό ε, κοινής αντιμετώπισης των κινδύνων. Πώς αυτή η ιδέα απαλήφθηκε από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για μια μελλοντική fiscal capacity. Και τέλος για την Ελλάδα για τις αποφάσεις που έχει λάβει η ομάδα Ευρώ, το Eurogroup παλαιότερα. Πότε νομίζετε ότι θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις αυτές από το πρόγραμμα δηλαδή της ε, αγοράς ασφαλιών στους ε, λογαριασμούς της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες που υπάγονται στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Επίσης, εδώ το κύριο χαρακτηριστικό πρέπει να είναι ότι πρέπει να είναι σημαντικού μεγέθους, δηλαδή ε, να έχουν, να έχουν σημασία. Μπορεί δηλαδή να μην είναι μεγάλες, αλλά μπορεί να αντιμετωπίζουν συστημικό κίνδυνο. Τότε με το κριτήριο αυτό μπορούν να μπουν ίσως στην ομάδα των 150. Είπαμε ότι είναι μεταξύ 130 και 150 τραπεζών. Θα εξαρτηθεί αυτό από διάφορα πράγματα μεταξύ άλλων και πόσες χώρες, αυτές που δεν έχουν ακόμη το ευρώ, θα ενταχθούν στο σύστημα. Τραπεζική ένωση χωρίς δημοσιονομική ένωση. Γνωρίζετε ότι η τραπεζική ένωση έχει τρεις πυλώνες, δύο από τους οποίους δεν προβλέπουν αμοιβαία αντιμετώπιση των κινδύνων. Ο τρίτος, ναι. Η κοινή εγγύηση των καταθέσεων δηλαδή. Το ζήτημα εδώ είναι ότι μπορείτε να έχετε τραπεζική ένωση σε ό,τι αφορά την εποπτεία και τους κανόνες και να διαρρήξετε τα δεσμά μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους κατά ένα βαθμό, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εποπτεία. Για να έχετε τότε την βεβαιότητα ότι ο κεντρικός επόπτης θα εξετάζει τράπεζες ανεξαρτήτως του που έχουν την έδρα τους ανεξάρτητα από τα εθνικά επενδυμένα συμφέροντα ή ενδεχόμενες εθνικές πολιτικές πιέσεις. Σε κάποιο βαθμό ο σύνδεσμος αυτός λοιπόν διαρριγνύεται. Ωστόσο, εάν πρέπει να επανακεφαλοποιήσετε μια τράπεζα που δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ESM, πάλι αυτό πηγαίνει στον εθνικό προπολογισμό. Έτσι λοιπόν διαρριγνύεται ο δεσμός μεν, αλλά όχι κατά 10%. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Όπως είπαμε όμως πολλές φορές, πριν να έχετε κοινή αντιμετώπιση των κινδύνων, πρέπει να αποδείξετε πρώτα ότι όλες οι χώρες επιθυμούν να μοιραστούν την κυριαρχία τους για τα δημοσιονομικά και ότι προτίθεται να εφαρμόσουν τους κανόνες τους οποίους οι ίδιες έχουν υιοθετήσει. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη και είναι, αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να δημιουργηθεί και μια κοινή ε, δημοσιονομική ένωση. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μοίρασε τα κέρδη SMB στις ε, τράπεζες, εθνικές τράπεζες, που δεν μπορώ να πω ότι διαπραγματεύονται, αλλά αναλόγως με τις εθνικές τους νομοθεσίες θα αποδώσουν ή και όχι τα κέρδη στις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες πάλι θα χρησιμοποιήσουν τα κέρδη αυτά για το πρόγραμμα, για την δημοσιονομική ικανότητα, fiscal capacity. Σε ό,τι αφορά να υπάρχει, δεν έχει, δεν έχει χαθεί και τελείως, γιατί γίνεται κάποια αναφορά στην δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθούν, να δημιουργηθούν μάλλον reform contracts. Και με τον τρόπο αυτό περιλήφθηκε τελικώς ε, αυτή η δημοσιονομική ικανότητα και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Τώρα, για το Λαϊκό Κόμμα Ο κύριος Φέιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις. Η, η πρώτη έχει να κάνει με το σύστημα και το κατά πόσο αυτό επιτυγχάνει τους στόχους λίματος και χρέους και που προβλέπονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη μαζί με ένα σύνολο κυρώσεων, αλλά νομίζω πως εκεί λείπει και ένα σύνολο κινήτρων. πολύς λόγος γίνεται για το σύστημα sticks και carrots αλλά νομίζω πως το δεύτερο το ξεχνάμε συχνά. Εμείς στην Πορτογαλία και στην Ελλανδία έχουμε προβλήματα και θα έπρεπε να υπάρξουν κίνητρα πέρα από το να μας λένε απλώς ότι είμαστε στον καλό δρόμο και ότι κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το δημόσιο χρέος. Σε πολλά κράτη αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, μη, έγινε λόγος για ταμείο εξαγοράς χρέους, για διάφορες άλλες λύσεις. Ο κ. Φάρομπόη προτείνει μια γενική λύση. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με αυτή την υπερβολική το υπερβολικό χρέος μέσα στα, νομικά, στα νόμιμα πλαίσια. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ευχηθώ καλές γιορτές, καλό 2013, καλύτερο από το 2012. Ήδη το Financial Times σας έβγαλε προσωπικότητα της χρονιάς που μας πέρασε. Έχετε λοιπόν μεγάλες, έχουμε μεγάλες προσδοκίες για τον επόμενο χρόνο από εσά. Σας ευχαριστώ. Ε, Δημοσιονομικέ προσαρμογέ έχω πει επανειλημμένω, ήταν αναπόφευκτες. Να μην ξεχάσουμε πώς στάσαμε σε αυτή την κατάσταση, καταρχήν. Δεύτερον, θα, υπάρχουν, ε, θα υπάρξει συρρήκνωση, φυσικά και θα υπάρξει. Βράχει πρόθεσμα. Πώς θα απαλύνουμε αυτά αυτέ τι επιπτώσει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένα, για παράδειγμα, είναι να εστιάσουμε περισσότερο στι δαπάνε, στη μείωση των δαπανών και όχι στι αυξήσει των φόρων. Δεύτερον, είναι να αναλάβουμε τι ε, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, ελπίζοντα ότι οι εξαγωγέ θα αυξηθούν. Έχουμε παραδείγματα χωρών που κατάφεραν να απαλύνουν τις επιπτώσει των αναπόφευκτων δημοσιονομικών διορθώσεων μέσω ψηλότερων εξαγωγών και αυτό θα πρέπει να έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτή είναι η στρατηγική κλειδί σε μια κατάσταση που ομολογουμένως είναι πολύ σοβαρή και πολύ οδυνηρή για αυτές τις χώρες. Οπότε, καθόλου ελαφριά την καρδία δεν εξετάζουμε αυτά τα, αυτές τις ανησυχίες. σε σχέση με τα υπερβολικά και εντυπωσιακά επίπεδα χρέους. Δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή γι' αυτά. Περισσότερες χώρες που είναι υποπίεση αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και η σημερινή στρατηγική στόχο έχει εν τέλει να μειώσει τα χρέη, σαν την αναλογία χρέους προς ΑΕΠ. Και θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ πολύ για τις χριστουγεννιάτικες ευχές σας και σας τις ανταποδίδω ολόψυχα σε όλους σας. Uh, ευχαριστώ. Προχωράμε στο Άλντε και στο Ραμόν Τρεμόσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα για τις προβλέψεις που μας παρουσιάσατε για την Ισπανία. Εκφράσατε την αισιοδοξία σας. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όλες οι προβλέψεις της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των διαφόρων Ισπανικών τραπεζών, αλλά και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αναφέρει ότι το 2014 θα είναι η χρονιά τεράστιας κρίσης στην Ισπανία. Θα αυξηθεί η ανεργία, θα μεγαλώσει, θα αυξηθεί το έλλειμμα, το χρέος, τα δημόσια οικονομικά θα εκτροχιαστούν πλήρως και θα δούμε και το ε, κόστος της ε, δημοσιονομικής διάσωσης τότε είναι που πραγματικά θα πληρώσουμε το τίμημα. Είπατε ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν πράγματι, αλλά αυτές αφορούν μόνο τρεις ή τέσσερις περιφέρειες. Η Καταλονία είναι υπεύθυνη για το 30% των ισπανικών εξαγωγών. Αυξήθηκαν οι εξαγωγές της Καταλωνίας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα μειώνεται αυτός ο ρυθμός αύξησης. Επιβραδύνονται μάλιστα οι εξαγωγές. Έχετε λόγους που πραγματικά υποστηρίζουν αυτή την ε, φιλοδοξία. Ευχαριστώ. Απάντηση. Οι προβλέψεις μου δεν αναφερόντουσαν στην Ισπανία, αναφερόντουσαν στο σύνολο της ζώνης του ευρώ και ως τέτοιες θα πρέπει να ερμηνευθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ραμόν Τρεμόσα πάλι. Να σας πω και το εξής. Περίπου πριν από ένα μήνα, ο Ισπανός Υπουργός Οικονομικών ήρθε εδώ στο Κοινοβούλιο και είπε λέξη προς λέξη η οικονομία της Ισπανίας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Ποια είναι η άποψή σας. Απάντηση του κυρίου Ντράγκη. Συγγνώμη αλλά δεν σχολιάζω τις δηλώσεις Υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών. Ωστόσο μπορώ να σχολιάσω τα γεγονότα και τα στοιχεία. Ε, και τα στοιχεία και τα γεγονότα δείχνουν ότι το πλεόνασμα των των τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε όταν μειώθηκε το μοναδίο κόστος εργασίας και άρα αυξήθηκαν και οι εξαγωγές. Υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις βελτίωσης. Είναι παθές, πιστεύω να μην παραδέχεται κανείς την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ισπανία, κάτι το οποίο ισχύει εν μέρη και για την Πορτογαλία και για την Ιρλανδία και για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες που δοκιμάζονται. Έχουμε σημειώσει οδυνηρή πρόοδο αυτή τη χρονιά και αυτό είναι αυτό που χαρακτηρίζει αυτή τη χρονιά. Ο κύριος Τρεμόσα. Έχω 1,5 λεπτό ακόμα. Όταν μιλάτε για το μοναδιαίο κόστος εργασίας, ε, ε, κάνετε το διαχωρισμό μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, διότι αν δεν απατώμε ο αντιπρόεδρος ο Ισπανός είπε ότι το δώρο των Χριστουγέννων ε, των Ισπανών δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο δεν κατεβλήθη φέτος, θα καταβληθεί του χρόνου. Και αυτές οι μειώσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας αναφέρονται μόνο σε και αφορούν πολύ λίγους υποτομείς του ιδιωτικού τομέα ο κύριος Ντράγκη. Όχι, το μοναδιακό κόστο εργασία αφορά στο σύνολο τη οικονομία. Από εκεί και πέρα όμω έχουν υπάρξει και μεταρρυθμίσει στην αγορά εργασία, και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω λοιπόν ότι η χρονιά αυτή χαρακτηρίζεται από οδυνηρή μεν πρόοδο, αλλά πρόοδο ούτω ή άλλω. Ευχαριστώ. Το ελπίζουμε, λέει ο κύριος ε, Τρέμοσα. Ο Ραμόν μας έδειξε ότι με σύντομες ερωτήσεις έχουμε και πολλές απαντήσεις από την πλευρά του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για το ΕΡΚ λοιπόν ο Ζων Πολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε ε, που βρίσκεστε εδώ μας εξηγήσατε με πολύ σαφείς όρους τους ε, διαφόρους οργανισμούς που θα δημιουργηθούν, θα συσταθούν, τις προθεσμίες, τη συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Εάν θυμηθώ τα λεγόμενα διαφόρων όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή εποπτεία προκειμένου να μετριάσουμε τις ελλείψεις του συστήματος οι οποίες διαπιστώθηκαν με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα ο στόχος που έχουμε θέσει είναι πολύ πιο μετριοπαθής και θέλω ε, πολύ ειλικρινά να σας ρωτήσω το εξής. Πώς ε, νομίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπέζα ότι θα τα καταφέρει καλύτερα από ό,τι τα έχει καταφέρει στο παρελθόν και ποια επιπρόσθετα μέσα θα έχει στη διάθεσή της για να φτάσει σε αυτό το σκόπο. Ο εξ μου θεωρεί ότι είναι ίσως ε, ερώτηση με κακία την οποία απευθύνω σε εσάς. Παραμονές Χριστουγέννου δεν θα έπρεπε. Αλλά πρέπει να την κάνω ούτως ή άλλως. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Είναι φυσικά τα ερωτήματα αυτά, ανακύπτουν φυσικά ε, και είναι καλό να προσπαθούμε να απαντούμε. Η απάντηση έγκυται στο γεγονός το εξής, ότι δεν νομίζουμε ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα από οποιαδήποτε εθνική εποπτική αρχή και ο λόγος είναι γιατί θα δουλέψουμε μαζί με την εκάστοτε εθνική εποπτική αρχή. Μαζί λοιπόν θα εφαρμοστούν αυτά και από εμά και από τις εθνικές αρχές. Το βασικό με αυτό το μηχανισμό εποπτείας είναι ότι θα υπερβούμε τα εθνικά σύνορα. Επομένως, θα υπερβούμε και αυτή την περιχαράκωση η οποία συνέβαλε στον κατακαιρματισμό της ζώνης του ευρώ. Και αυτή είναι και η απάντηση που έδινα πάντοτε. Δεν είχα ποτέ καμία φιλοδοξία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ποτέ δεν θεωρούσα ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα ή τουλάχιστον ποτέ δεν το θεωρούσα και το δήλωσα πριν αυτό να συμβεί και πριν πραγματικά να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Πίτερ Σκίνερα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν λέω ότι είστε υπερήρωας, αλλά σίγουρα είστε ο καλύτερος άνθρωπος από τον κόσμο της οικονομίας ε, αυτή τη χρονιά, λόγω των δυσκολιών που έχετε αντιμετωπίσει. Ξέρουμε βέβαια τώρα ότι ο αριθμός των τραπεζών που θα εποπτευθούν άμεσα από τον μηχανισμό εποπτείας είναι 150. Έρετε, έχετε όμως στοιχεία για το πόσες τράπεζες ενδεχομένως μπορούν να μπουν σε αυτό το ε, εργαλείο για την άμεση ανακεφαλοποίησή τους. Ε, υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα προς το θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προβούμε τώρα σε τέτοια εκτίμηση, γιατί είναι διαφορετικές ε, οι διαδικασίες. Γνωρίζουμε ποιες τράπεζες ενδέχεται να το ζητήσουν επειδή έχουν την έδρα τους σε ορισμένες χώρες και υπάγονται στον, στη διαδικασία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Αλλά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ποιες χώρες θα χρειαστούν άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον σταθεροποιητικό μηχανισμό. Αυτός ο ίδιος ο μηχανισμός θα πρέπει να το κρίνει αυτό, ο ESM δηλαδή ο ESM θα χρησιμοποιήσει την εποπτεία του άλλου μηχανισμού, του ενοποιημένου μηχανισμού εποπτείας του SSM ως στήριξη για τη λήψη αποφάσεων του. Αλλά ο ESM είναι εκείνο ο μηχανισμός ο οποίος τελικά θα αποφασίσει. Άρα στην πράξη είναι δύσκολο, αλλά στη θεωρία ίσως είναι δυνατόν να γίνει εκτίμηση αυτή. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Για τη γενική οικονομία αφενός υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος του υψηλού πληθωρισμού και αφενός υψηλής ανεργίας, και αφετέρου της υψηλής ανεργίας. θέλετε να διαχωριστούν οι πολιτικές και θεωρείτε ότι μια και τώρα είναι Χριστούγεννα και έρχεται και ο Άγιος Βασίλης, αναμένουν πολλά από εσά ω όθηση για τι οικονομίε του οι διάφορε χώρε μέλη. Μήπω θα είστε εσεί όμω τελικά ο Τσιγκούνης Κρούντζ, ο οποίος ε, τις περιμένει στη γωνία. Κύριος Δράγκη, φέτος, όπως είπα και πριν, κάναμε δύο ε, operations μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότηση ε, με ασφάλεια. Δεν είναι το καλύτερο εργαλείο για να δώσει χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση για δανειοδοτήσεις. Διότι εφόσον δανειοδοτούν οι τράπεζες παράγουν και ασφάλεια την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δανειοδοτηθούν από εμά. Τα επιτόκια είναι χαμηλά. Τα πραγματικά επιτόκια είναι και αρνητικά σε πολλά σημεία της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα έχει διατηρηθεί, έχει εξασφαλιστεί η σταθερότητα τιμών και μέσω και μακροπρόθεσμα οι προβλέψει για τον πληθωρισμό αυτό δείχνουν ότι θα είναι σταθερέ τιμέ. Νομίζω ότι αυτά καταφέραμε φέτο. Και αυτά θα μείνουν μαζί μας και είμαστε αρκετά πεπισμένοι ότι αυτή η νομισματική μας πολιτική στέκεται στα πόδια της και με τον καιρό θα παραγάγει μια καλύτερη οικονομική κατάσταση από αυτήν που βλέπουμε σήμερα. Μάλιστα για τον λόγο αυτό η πρόγνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μάλλον οι προβολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προβλέπουν ε, ε, αρχή ανακάμψεως για το, εξάμεινο το, επόμενο, το δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους. Ο Πίτερ Σκίνερ τελείωσε. Ο Γκέι Μίτσελ. Ε, ε, ε ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω και με άλλους συναδέλφους και θα ευχηθώ στον κύριο Τράγκη καλά Χριστούγεννα και ελπίζω να, να πάνε καλά. Ελπίζω ότι στις 17 Μαρτίου του Αγίου Πατρικίου οι Ιρλανδοί να έχουν λόγο να χαμογελούν και πάλι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την αναδιάθρωση του αγγλοϊρλανδικού χρέου. Αλλά δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Πολλοί μα λένε και κυρίω κάποιοι οπορτουνιστέ, ότι η λιτότητα δεν, χρησιμοποιεί, δεν, ε, δεν αποδίδει. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο χρησιμοποιεί σήμερα και αύριο ή σε μια χαρά. Ταυτόχρονα όμω, θα χάσουμε την υποστήριξη του κοινού, του κόσμου, αν δεν του προσφέρουμε κάποια ελπίδα. Γι' αυτό ρωτώ κύριε Ντράκη το εξή ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, κύριο Σόιπλε, γράφοντας στο Wall Street Journal την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε στον Χόλκετ Σνάιντερ της Μπάρνμπεργκ στο Λονδίνο και πρόσφατη ανάλυση του Συμβουλίου της Λισαβόνας και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μείνει στο μονοπάτι αυτό μπορεί να εμφανιστεί εν τέλει η πιο σημαντική η πιο ζωντανή οικονομία του δυτικού κόσμου. Συμφωνεί ο πρόεδρος Τράγκη με αυτή την ε, τοποθέτηση. Ναι, συμφωνώ με την άποψη αυτή, διότι η Ευρωζώνη έχει κατά κάποιο τρόπο τα καλύτερα θεμέλια που μπορεί να βρει κανείς σήμερα. Αν εξετάσετε τα δημοσιονομικά ελλείμματα, χρέος ε, τρεχόντων ε, λογαριασμών, τιμές, πληθωρισμό. Όποια, όποια παράμετρο και να εξετάσετε, θα βρείτε μια λιγότερη, μια μικρότερη έλλειψη ισορροπίας από σχεδόν τα περισσότερα άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό που πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε είναι να βασιστούμε, να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα γερά θεμέλια ως Ευρωζώνη, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό μας που κατά κάποιο τρόπο απομονώνει τις χώρες και τις καθιστά έγκλειστες στις ε, δικές τους αδυναμίες. Αυτή είναι η πρόκληση. Και φαίνεται ότι φέτος τουλάχιστον προχωρήσαμε αρκετά προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του στόχου. Στην διόρθωση δηλαδή των ανισορροπιών και δημοσιονομικών και διαφθορτικών και από άποψη ανταγωνιστικότητας αλλά και στο επίπεδο της διαχείρισης της διακυβέρνησης δηλαδή, ώστε να φτιάξουμε μια πιο σκόπιμη, πιο γνήσια νομισματική ένωση. Ας μην λησμονούμε όταν εξετάζουμε τις θεμελιώδεις μας αυτές, τις, ε, τις βάσεις μας αυτές, τα θεμέλια μας αυτά, είναι γενικώ καλά και προσφέρουν μια καλή βάση για το σχόλιο που έκανε άλλωστε και ο υπουργό κ. Σόιπλε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτό το θετικό χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Ωστόσο είναι σημαντικό να πω ότι λέμε διαρκώς στον κόσμο τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν τους λέμε γιατί. Εγώ θα έλεγα και στο δικό σας επίπεδο ως Προέδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έχετε κάνει καλή δουλειά και θα έπρεπε να σας το λέμε και περισσότερο, αλλά στο δικό σας επίπεδο και στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να αρχίσουμε να εξηγούμε περισσότερο το γιατί. Να αρχίσει ο κόσμος να καταλάβει ότι υπάρχει και κάποια ελπίδα, δηλαδή το κάνουμε για κάποιο σκοπό. Ας γίνει λοιπόν αυτό περισσότερο το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουμε το 2013. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις σας. Ο κύριος Δράγκη, ευχαριστώ πολύ, ιδίω και για την πρότασή σας, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο επεξηγηματικοί στα σχόλιά μας και στο τι εξηγούμε στον κόσμο. Ε, σίγουρα εγώ θα το σημειώσω και θα το υιοθετήσω. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται ο νομισματικός διάλογος. Ο επόμενος έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δευτέρου του 2013. Μην σηκωθείτε να φύγετε όμως όλοι, διότι έρχεται ο Υπουργός κύριος Σιαρλής στο τέλος της Κυπριακής Προεδρίας ε, και αυτό, δηλαδή θα προσέλθει εδώ στις 5 ε, και μισή. Πάντως, για όσους και όσες φεύγετε, θυμηθείτε ότι αύριο δεν συναντώμεθα εδώ, αλλά στην αίθουσα 2Q2, γιατί εδώ θα συνεδριάσουν οι πρόεδροι ομάδων. Θα συνεχίσουμε σε 5 λεπτά. Okay, we now, uh, Είμαστε έτοιμοι. Για το επόμενο μας σημείο, που είναι η ανταλλαγή απόψεων και ο οικονομικός διάλογος με τον εκπρόσωπο και προεδρεύοντα του Συμβουλίου Εκοφήν, κύριο Βάσιο Σαρλή. Θα του δώσω το λόγο στον κύριο Σαρλή για 10 λεπτά και έπειτα θα έχουμε 5 λεπτή ερωταπάντηση για καθέναν. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, I would like to begin with... Ναι, ναι. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω με την εξή δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει η μεγαλύτερη ενιαία αγορά και το ευρώ παραμένει ισχυρό νόμισμα ακόμα και σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΑ, και τις ε, μακροοικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν το περασμένο μήνα, οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, συρρυκνώνονται κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του χρόνου. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση σημαίνει ισχνές προπτικές για αντιστραφή της μεγάλης αύξησης στην ανεργία, ιδιαίτερα ανεργία των νέων, αύξηση της ανεργίας που έχουμε εδώ και τρία χρόνια. Αυτή η ανεργία είναι ένα από τα, τις πιο ανησυχητικές πτυχές της ε, σοβούσας ε, οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεχιζόμενη κρίση στο Ευρωζώνη έχει αρνητικέ επιπτώσει στην εμπιστοσύνη, την επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Παγκοσμίω η έλλειψη εμπιστοσύνη πλήττει περισσότερο την Ευρωζώνη των 17, γι' αυτό πρέπει να βρεθούν βιώσιμες λύσεις για την κρίση. Αν και πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν εφαρμόσει σημαντικές διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, παραμένουν αρκετές προκλήσεις που πρέπει να ακόμα να αντιμετωπιστούν. Ε, όλοι γνωρίζουμε πως τα κέρδη από τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις ε, είναι μεγάλα και κυρίως ε, προκύπτουν μέσω πρόθεσμα και επηρεάζουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Τέλος, η επίλυση των τραπεζικών προβλημάτων της Ευρωζώνης ώστε να δημιουργηθούν αξιόπιστες αγορές, η e ευφυής δημοσιονομική εξυγίανση ε, φαίνεται να είναι κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα να σας περιγράψω τα τελευταία από συμπεράσματα του Συμβουλίου της περισμένης εβδομάδας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για έναν οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της ΟΝΕ επί τη βάση βαθύτερης ολοκλήρωσης και ενίσχυσης της αλληλεγγύης. Είναι ε, επιτακτική ανάγκη να σπάσει ο φαύλος Κύκλο ανάμεσα στι τράπεζε και τα δημόσιο, τα κρατικά χρέη. Μετά από τις δηλώσεις του Ιουνίου και Οκτωβρίου 2012 θα πρέπει σύντομα να συμφωνηθεί ένα νέο πλαίσιο στο πρώτο εξάμεινο του 2013, έτσι ώστε όταν θα συσπιστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός εποπτείας, θα έχει, να έχει τη δυνατότητα να ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες άμεσα. Στο πλαίσιο που η τραπεζική εποπτεία θα κινηθεί αποτελεσματικά προς έναν ενιαίο υποπτικό μηχανισμό, ε, θα απαιτηθεί και ένας ενιαίος μηχανισμός διάλυσης εξαγοράς τραπεζών. Γι' αυτό η Κομισιόν θα υποβάλει το 2013 μια πρόταση για έναν ενιαίο μηχανισμό ε, διάλυσης τραπεζών για τα μέλη που συμμετέχουν στον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό που θα εξεταστεί ως θέμα προτεραιότητας με στόχο να υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια, ε, να υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την διάλυση χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων, ενώ θα προστατεύονται οι φορολογούμενοι στο πλαίσιο δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Για να εξασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, καθώ και να αυξηθεί η επασχόληση, κυρίω στην Ευρωζώνη αλλά και σε ολόκληρη την Ένωση, διάφορα άλλα ε, θέματα θα εξεταστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2013. Τα θέματα αυτά αφορούν το συντονισμό των εθνικών προγραμμάτων, την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, την σκοπιμότητα και τον τρόπο εφαρμογής αμοιβαία υπεφωνημένων συμβάσεων για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και τους μηχανισμούς αλληλεγγύης και μέτρα για να προωθηθεί η εμβάθυνση της νέας αγοράς και να προστατευτεί η ακυρεότητά της. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η δημοκρατική νομιμότητα και η λογοδοσία θα εξασφαλιστούν περαιτέρω ολοκλήρωση της άσκησης πολιτικής και μεγαλύτερη συγκέντρωση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής και εμπλοκής του Ευρωκοινοβουλίου. Διαδικασία που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της δημιουργίας νέων μηχανισμών που θα αυξήσουν το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στο εθνικό, στα εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση καθώς και με βάση το πρωτόκολλο υπαρθμών 1 συνθήκων. Το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα καθορίσουν από κοινού την οργάνωση και την προώθηση μιας διάσκεψης των εκπροσώπων τους για να συζητηθούν τα θέματα τα σχετικά με την ΟΝΕ για την Ελλάδα. Το Eurogroup και κατά συνέπεια το Συμβούλιο πρόσφατα συμφώνησαν για τροποποίηση του της δημοσιονομικής προσαρμογής καθώς και να παρατείνουν την προθεσμία για τη διόρθωση του χρέους μέχρι το 2016 και μαζί με τις ελληνικές αρχές συμφώνησαν για μέτρα για αντιμετώπιση της ε, κρίσης καθώς και μείωση του χρέους μέχρι το 2016 και το 2020 στο 124% του ΑΕΠ. Ε, καλωσορίζουμε τις πρόσφατες αυτές εξελίξεις καθώς και τη θετική ε, αντίκτυση της, ε, το θετικό αντίκτυπο της ε, επαναγοράς των, του χρέους. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τη διαπραγματευτική ομάδα για τη σπουδαία τους προσπάθεια και την αίσθηση συμβιβασμού, το πνεύμα συμβιβασμού που μας επέτρεψε σχεδόν να κλείσουμε το θέμα. Το θέμα Γκοζές έχει κλείσει και όλα τα σημεία έχουν συμφωνηθεί. Στην έκθεση Φερέρα υπάρχει ένα σημείο που εκκρεμεί. Γερήτρα αναθεώρησης και σε σχέση με αυτήν η δήλωση της Κομισιόν για τον οδικό χάρτη για την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Τα προτιμούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει και σε αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κοινή βάση για θέματα όπως τα ευρωμόλογα ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξαγοράς Χρέους. Υπάρχουν όμως και νομικές, ε, νομικοί προβληματισμοί σε σχέση με το τι είναι εφικτό επί τη βάση της ισχύουσα συνθήκης και τι όχι. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο της περισμένης εβδομάδας συμπέρανε πως χρειάζεται περισσότερη δουλειά για αυτό το θέμα και άρα το πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνεργασία συνεργασία με τον πρόεδρο της Κομισιόν και σε διαβούλευση με τα κράτη-μέλη θα υποβάλει στον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2013 πιθανά μέτρα, καθώς και ένα δεσμευτικό χρονικά οδικό χάρτη για διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού αλληλεγγύης. Θα ήταν πρόημο να συμπεράνουμε κάτι για αυτές τις νομοθεσίες που θα προκαταλαμβάνοντας τα πορίσματα αυτών των, την έκφαση μάλλον αυτών των επιπλέον διαπραγματεύσεων που πρέπει να γίνουν. Ελπίζω πως το σχέδιο της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου μαζί με τη δέσμευση της Κομισιόν για έκδοση δήλωσης θα μας ε, βρουν απόλυτα σύμφωνος. Επίσης ε, ελπίζω πραγματικά πως θα μπορέσουμε για μια ακόμη φορά να αποδείξουμε πως η κοινοτική μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει για τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτόν. Όπως όλοι γνωρίζετε, η συμφωνία που επετεύθη κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εκοφήν την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν εύκολη. Μετά από 15 ώρες συνεδρίας και την... τα πολλά και διάφορα θέματα που χρειαζόταν να εξετάσουμε. Η συμφωνία σέβεται τις πέντε βασικές αρχές που θέσπισε το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο, με συγχωρείτε. Σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην νομισματική πολιτική και τις εποπτικές λειτουργίες στην ΕΚΤ. Ισότιμη μεταχείριση κατών μελών εντός ή εκτός ευρωζώνης που συμμετέχουν στο μηχανισμό. Τρίτον, κατάλληλα μέτρα λογοδοσίας. Τέταρτον, το ο νέος μηχανισμός θα ε, βασίζεται στα υψηλότερα στάνταρ για την εποπτεία την τραπεζική και η ΕΚΤ θα εποπτεύει τα διάφορα πιστοτικά ιδρύματα με διαφοροποιημένο τρόπο ενώ θα κάνει αυξημένο έλεγχο των πιο μεγάλων τραπεζών στα κράτη-μέλη. Πέμπτη αρχή ήταν μια αποδεκτή και ισορροπημένη λύση για τον τρόπο ψηφοφορίας και τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Για το Συμβούλιο ήταν πολύ σημαντικό η ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς να γίνει απόλυτα σεβαστή στη δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Επίσης ήταν σημαντικό να εξασφαλιστεί πως η δημιουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού δεν θα μεταβάλει την ισορροπία των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Εθνική Αρμοδιαρχή και την ε, Ευρωπαϊκή ε, Τραπεζική Αρχή. Αφού τώρα αυτά όλα έχουν ξεκαθαριστεί, μπορούμε από κοινού να οριστικοποιήσουμε το προβλεπόμενο υποπτικό πλαίσιο. Είμαι πεπισμένο ότι είμαι σίγουρο ότι οι επερχόμενε διαπραγματεύσει για τον υποπτικό μηχανισμό θα οδηγήσουν σε συμφωνία για την υποπτία των τραπεζών με βάση τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές. Υπό το φως των εξελίξεων των τελευταίων ετών όλοι συμφωνούμε πως αυτό είναι πολύ σημαντικό CRD4. Ε, σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου προχωρήσαμε για, την, ε, για ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και η οδηγία CRD4 Κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας της Κύπρου, από κοινού κάναμε σημαντική πρόοδο για αυτή γι' αυτό το νομοθετικό πακέτο. Οι μελλοντικέ διαπραγματεύσει τώρα θα εστιάσουν μόνο σε ένα περιορισμένο αριθμό κρεμών ζητημάτων. Η συμφωνία αυτή είναι δυνατή, αλλά πρέπει ακόμα να δουλέψουμε από αυτής. Σήμερα δεν θα σχολιάσω με λεπτομέρειες κανένα από τα εκκρεμή ζητήματα. Το κατάλληλο σημείο, κατάλληλο βήμα μάλλον, είναι ο τριμερής διάλογος. να τονίσω και πάλι και ίσως θα έπρεπε ακόμα και να δεσμευτώ και να ζητήσω από τους Ιρλανδού Ιρλανδούς συναδέλφους, γιατί είναι ένας, ένα θέμα όπου το Συμβούλιο αποδίδει ψηλή προτεραιότητα και είμαι βέβαιος πως και εκείνοι θα το κάνουν. Θα θυμίσω πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13 και 14 Δεκεμβρίου επανέλαβε τη σημασία κανόνων για το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και ζήτησε ταχεία υιοθέτηση για την CRA3 να σας ε, πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί καταφέραμε πολιτική συμφωνία για τις, ε, τους οργανισμούς πιστοληπτικής ε, δυνατότητας, αξιολόγησης, με συγχωρείτε θέλουμε να υπάρχει ένα πολύ πιο στεναρό και υγιές περιβάλλον για την χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Μειώθηκε η αυτόματη εξάρτηση από τις αξιολογήσεις καθώς και ε, έγινε λόγος για την ευθύνη των ε, των οργανισμών αυτών. Σημαίνει αυτό διαφάνεια στους κανόνες καθώς και μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τις αξιολογήσεις αυτές στις αγορές. Τέλος. Ε, καλωσορίζω την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωκοινοβούλιο για τα κεφάλαια κινδύνου και για τα κοινωνικά ταμεία. Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, εξ ονόματο τη Κυπριακή Προεδρία θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την μόνιμη προσοχή που δίνει στο θέμα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Γνωρίζω το μεγάλο και μόνιμο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Ε, επίσης θα πρέπει να αναφέρω από την έκθεση της κυρίας Ποδηματά ε, επί ενός κοινού συστήματος για τη φορολόγηση των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που υιοθετήθηκε φέτος το Μάιο καθώς και το νομοθετικό ψήφισμα που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο το Συμβούλιο έστρωσε τον δρόμο για μια διαδικασία αυξημένη συνεργασία που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη που έχουν δείξει μεγάλη στήριξη στην αρχή της εισήγηση ε, ενό τέτοιου φόρου να προχωρήσουν μόνα τους. 11 κράτη-μέλη επέλεξαν να μπουν στην ε, ισχυμένη συνεργασία σε αυτό το στάδιο και ακόμα ένα ε, εξετάζει το ενδεχόμενο. Γι' αυτό η Κομισιόν έχει υποβάλει πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για, την, να, για να εγκριθεί η αυξημένη συνεργασία. Η Προεδρία δούλεψε πολύ στην εξέταση αυτών των προτάσεων και είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο ε, γιατί εξετάσαμε το θέμα και δόθηκε τελικά η έγκριση για την, ε, την ε, αυξημένη συνεργασία από πλευρά του Κοινοβουλίου. Τώρα το Συμβούλιο πρέπει να ολοκληρώσει τις συζητήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ επίσης διότι έχω εδώ ένα σημείωμα, μια συνοπτική ε, έκδοση των σημειωμάτων της, ε, της Προεδρίας έχετε λάβει υπόψη σας την έκθεση Γκοζές λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περιλάβει τις απόψεις του για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, και στις 26 Οκτωβρίου 2012. Σας ευχαριστώ λοιπόν που σημειώσατε εδώ τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις και ίσως το καλύτερο είναι να αρχίσει το Λαϊκό Κόμμα με τον Ζαν Πολ Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είμαστε μεταξύ μας λίγο πολύ απόψε και ας μιλήσουμε απλά. Ακόμη και αν δεν υπάρχει μεγάλο πλήθος ευρωβουλευτών, ωστόσο είναι παρόντες όσοι συνεργάστηκαν με την Κυπριακή Προεδρία. Κάτι που δείχνει ότι ήταν σημαντική η εντύπωση που άφησε η Κυπριακή Προεδρία γιατί είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Δεύτερο, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι όπως και ο Λανάρντο ο οποίος θα πει και αυτός ε, λίγα λόγια γιατί ήταν ε, γιατί έχουμε το δεύτερο ε, κείμενο για τους οίκους ε, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και για, το, για τη δέσμη των δύο μέτρων, όπως είπατε και εσείς, έχουν προχωρήσει τα πράγματα και για μας έχουν ολοκληρωθεί και εσείς και οι συνεργάτες σας μετά από μια περίοδο δοκιμών, να το πω έτσι, γιατί όπως είπα θα μιλήσουμε ειλικρινά, από μια περίοδο κάπως δύσκολη έναρξης, γιατί χρειάστηκε και εσείς να συνηθίσετε στο τι σημαίνει προεδρία και μάλιστα σε περίοδο ε, κρίσεως, με δυσκολίες για να συμβάλλετε στην, στο να συμφωνήσουν οι χώρες μέλη. Βέβαια ήταν όπως είπα μια αρχή κάπως δύσκολη, μετά τα πράγματα διορθώθηκαν και ε, δόθηκε, ε, επιτεύχθηκε μια επιτάχυνση ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο φάκελο αυτό αλλά και σε άλλους. Δεν θα σας θέσω ερώτημα τόσο πολύ για το μέλλον. Εσείς εξηγήσατε τι, τα, ποια είναι τα πράγματα μας περιμένουν. Είπατε ποιες είναι και οι αποφάσεις του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο δίδαγμα αντλείτε εσείς από την Κυπριακή Προεδρία και πώς θα προσπαθήσετε τα χρόνια που έρχονται να εξηγήσετε στις χώρες μέλη τι σημαίνει μια πραγματική διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι οι συνεργάτες σας κατανόησαν μέσα από τις συζητήσεις μας ότι η συναπόφαση δεν ε, ήταν ε, απλώς μια ακρόαση από πλευρά του, κοινοβουλίου των απόψεων, του, ε, του Συμβουλίου των Απόψεων του Κοινοβουλίου, αλλά μια πραγματική διαπραγμάτευση όπου δεν είναι πρόκειτο απλώς και μόνο για ευγενική ακρόαση των μένα από τους δε, αλλά για μια προσπάθεια αλληλοκατανόησης. Γι' αυτό και ρωτώ ε, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας και αν προτίθεστε στο μέλλον στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου να αναφερθείτε στην εμπειρία αυτή της Κυπριακής Προεδρίας ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει μεταξύ των δύο οργάνων, του Συμβουλίου δηλαδή Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ και εσά και τους συνεργάτες σας. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θέλετε να απαντήσετε. Μήπω θα θέλατε να ομαδοποιήσουμε τι ερωτήσει ή να απαντήσω αμέσω στον κύριο Κοζέση. Έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο για να κάνουμε ερωτήσεις-απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τα θετικά σας σχόλια, για την πρόοδο που επιτύχαμε και ιδίως για τους φακέλους που μπορέσαμε να κλείσουμε. Σημαντικό νομίζω είναι εδώ να υπό ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, είσαστε και εσείς και εμείς που με συνεργασία καταφέραμε να κλείσουμε τα θέματα. Και το δίδαγμα που αντλώ είναι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με τον τρόπο αυτό. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος πρόοδου, δηλαδή με συνεργασία. Και νομίζω ότι, ότι όπως ξεκινήσαμε, η απογείωση ήταν λίγο ανώμαλη, ας το πω έτσι, όπως εξήγησατε κι εσείς. Μέσα στη διαδικασία ωστόσο βρήκαμε τα πατήματά μας και καταλαβαμε ότι συνομιλώντας, ότι διαπραγματευόμενοι με γνώμονα το κοινό καλό, το καλό της Ευρώπης δηλαδή, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Και όλοι οι φάκελοι που παραμένουν ανοιχτοί και που θα αναλάβει την εκπαίδευσή τους η επόμενη Ιρλανδική Προεδρία, νομίζω ότι από αυτόν θα συνεχίσουν το έργο που αρχίσαμε εμείς. Και βεβαίως εκείνο που αναλάβαμε εμείς από την Ιδανική Προεδρία και ούτω καθεξής. είναι ο ρόλος που ε, καλούμαστε να παίξουμε. Όλα για την Ευρώπη. Εάν κοιτάξουμε προς τα πίσω, αυτό, είναι, αυτό επιτύχαμε. Κάθε τι που προσπάθησε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με επιμονή και επιμονή, επιτεύχθηκε τελικά. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις όπου ίσως να βιαστήκαμε υπερβολικά, ίσως επειδή ήταν απαραίτητο να γίνει γρήγορα. Και χαίρομαι πάντως που μπορώ να πω ότι για παράδειγμα ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που βασικά ήταν ένα εγχείρημα που προωθήθηκε μέσα σε έξι μήνες κατέληξε σε αίσιο πέρας γιατί ήταν σωστό για την Ευρώπη, ουσιώδες για την Ευρώπη και η συνεργασία που δεχτήκαμε από τις χώρες μέλη είχε το καλό αυτό αποτέλεσμα που όλοι επένεσαν την προηγούμενη εβδομάδα μετά από μαραθώνια συνεδρίαση και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο βήμα θα αποδειχθεί το ίδιο επιτυχές στις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα το δίδαγμα είναι ότι όλοι πρέπει να συνομιλούμε και να διαπραγματευόμαστε. Η συνθήκη της Λισαβόνας και η συναπόφαση δεν ήταν ισμάτιν Νομίζω ότι κάναμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο και αυτός είναι ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρο. Ευχαριστώ η κυρία Ελίσα Φερέιρα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα τα πω στα αγγλικά καλύτερα, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για όλους. Σας ευχαριστώ για την εργασία που καταβάλατε. Ε, Ιδίω εγώ συμμετέσχω στην επεξεργασία του λεγόμενου two-pack της δέσμης των δύο μέτρων και συμφωνώ με τον κύριο Γκοζές και σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για την εργασία σας, για την υπομονή σας. Ευχαριστώ και το προσωπικό σας, διότι πράγματι επιτελέσαμε πρόοδο. Νομίζω ότι αυτό που ελπίζαμε, δηλαδή να κλείσουμε τον φάκελο στη διάρκεια της δικής σας προεδρίας και αν δεν το επιτύχουμε, και έστω και αν δεν το επιτύχαμε, σχεδόν το επιτύχαμε, μένουν κάποιες τελικές προσαρμογές όπου θα θέλαμε κάποιες αιτιολογικές σκέψεις και κάποιες ε, ρήτρε επανεξέτασης που θα θέλαμε να δούμε να αρχίζουν με δήλωση της ε, Κομισιόν, όχι για να κάνουμε παράλογα πράγματα, αλλά τουλάχιστον έχουμε την εγγύηση ότι ορισμένα θέματα όπως πώς να διαχειριστούμε τα αποθέματα που έχουν συγκεντρώσει οι μέλη, ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν, ότι θα αναζητηθεί λύση και όχι ότι θα παραγωνιστούν. Μαζί επίσης και με τη δική μας αξίωση, ορισμένοι δηλαδή μηχανισμοί να βοηθήσουν τις χώρες να αντισταθμίσουν τις αρνητικές πτυχές του οικονομικού δυναμισμού και να υπάρξουν ορισμένα στοιχεία τα οποία να οδηγήσουν σε κάποια ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Και πάλι σας ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί σας στο ότι επιτύχαμε πρόοδο και τώρα που βρισκόμαστε στην τελική φάση της Προεδρίας σας και που πιθανόν είστε και πιο ελεύθερος να προβείτε σε έναν απολογισμό. Θα έρθω σε αυτό το πρώτο πράγμα που ε, αναφέρατε στην εισήγησή σας. Ένα ε, θεμελιώδες ερώτημα. Πώς εσείς δηλαδή στο ΕΚΟΦΗΝ αντιμετωπίζετε όχι την ανάγκη διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν συνιστάτε και μιλούμε για μέσα στο εξάμεινο, μια νέα διαδικασία δηλαδή, όπου κάνετε συστάσεις στις χώρες μέλη, οι συστάσει αυτές εφόσον δεν ακολουθηθούν από τις χώρες, οι χώρες αυτές θα βρεθούν σε δυσκολία τότε και υπάρχει μάλιστα και πρόβλεψη κυρώσεων, ποια είναι η εσωτερική αντίδραση του ΕΚΟΦΗΝ όταν βλέπετε ότι όλες οι προγνώσεις που κάνετε σε σχέση με τις συστάσεις σας αυτές μετά ανατρέπονται από τα γεγονότα. Για παράδειγμα, νούμερα. Ελλάδα. Ένα χρόνο πριν, 2011, η εκτίμηση για ανάπτυξη ήταν 0,7%. Τον ίδιο χρόνο κατέληξε στο μείον 6,9%. Για το 2012 η πρόγνωση ήταν 1,1. Καταλήξαμε ή καταλήγουμε μείον 6. Πορτογαλία, η οποία ακολούθησε τη συνταγή, η πρόγνωση για το 2011 ήταν αύξηση 0,7%. Η τελική έκβαση ήταν μείον 1,7%. Για το 2012, φέτος δηλαδή, η πρόγνωση ήταν συν 0,8%. Η τελική έκβαση μάλλον θα είναι 3,3 μείον. Για την Ευρωζώνη είχαμε μια πρόγνωση ανάπτυξη φέτο 0,5%. Θετική 0,5%. Τώρα καταλήγουμε στο μείον 0,4%. Όταν αντιμετωπίζετε λοιπόν χώρες οι οποίες ακολούθησαν τη συνταγή και παρέχομαι πάλι σε αυτό το εξάμεινο, συστάσεις προς τις χώρες και μιλώ για συγκεκριμένες χώρες, αλλά αυτό ισχύει για όλους εν τέλει. Μας λέτε, ακολουθήστε τη συνταγή, θα σας επιβάλλουμε κυρώσεις εάν δεν την ακολουθήσετε. Όμως επανεξετάζετε την ποιότητα των ε, συστάσεων που κάνετε και δεν απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά βέβαια, αλλά στο Συμβούλιο, στη, από την εμπειρία σας στο ΕΚΟΦΗΝ. Τίθεται το θέμα αυτό μέσα στο ΕΚΟΦΗΝ. Κοιτάτε λίγο και αυτά τα νούμερα, εξετάζετε για ποιο λόγο άραγε δεν επέτυχαν. Δεν επέτυχαν. Κάνετε κάτι αναμένοντας ένα αποτέλεσμα. Και βλέπετε ότι το αποτέλεσμα είναι τρει και τέσσερι φορέ αρνητικότερο από αυτό που είχατε προβλέψει. Είναι μεγάλο το θέμα. Δεν μπορείτε να ζητάτε θυσίε, σοβαρέ θυσίε από του πολίτε. να κάνουν τι θυσίε αυτές για να επιτύχουν κάποιο αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα αυτό δεν έρχεται ποτέ πολιτικά. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή εδώ όπως είπαμε κάπως είμαστε σε στενό οικογενειακό κύκλο, θα θέλαμε να καταλάβουμε με ποιο τρόπο δέχεται τα μηνύματα αυτά το ΕΚΟΦΗΝ και ε, ποια είναι η λογική που ακολουθεί στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ για τις ευθείες και ακαλόπιστες ερωτήσεις σας. Έχετε δίκιο. Για όλα όσα είπατε είναι σχεδόν, πώς να πω, ντροπή να κάνει κανείς προγνώσεις και να πετυχαίνει αποτελέσματα που είναι τόσο έξω από τις προγνώσεις αυτές. Από την άλλη μεριά, εξετάζοντας το, αυτό απηχεί την αστάθεια της κατάστασης που διερχόμαστε αυτή τη στιγμή. Και αυτό ενισχύει μάλλον το ρόλο που παίζουμε όλοι μας και Κομισιόν και Συμβούλιο και Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τρόπο σοβαρό αλλά και ταχύ, έτσι ώστε να βρούμε τι απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα. Όντω ε, αισθάνεται κανεί αμήχανα όταν βλέπει τι αποκλήσει αυτέ από, τις, ε, σχεδόν θετικέ προγνώσει τι οποίε αναμέναμε να επαληθευτούν και να, έχει, να έχουμε εν τέλει τόσο αρνητικά αποτελέσματα. Η σύντομη εμπειρία μου ε, τη ε, Προεδρία μου του ΕΚΟΦΗΝ με διδάσκει ένα πράγμα. Εάν 27 Υπουργοί Οικονομικών μπορούν να καθίσουν μαζί και να αντιμετωπίσουν, να συζητήσουν τα θέματα αυτά, είμαι πεπισμένος ότι εν τέλει θα βρουν τη λύση. Αν έγιναν λάθη, και πολύ πιθανόν να έγιναν, να έγιναν λάθη στην διαδικασία, στην πορεία, είναι λάθη που μπορούν να διορθωθούν προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών καθώς προχωρεί ο χρόνος. Και να δεχθούμε ότι για παράδειγμα έγινε ένα λάθος, ότι έγινε δηλαδή μια πρόγνωση ότι θα υπάρξει μια ανάπτυξη της τάξης του 0,2% και εν τέλει καταλήγουμε σε ένα έλλειμμα 1 ή 2% είναι άσχημο. Νομίζω όμως ότι διδασκόμαστε από τη διαδικασία αυτή. Και κάτι που μάθαμε, ένα από τα πολλά μαθήματα δηλαδή που ε, διδαχτήκαμε, είναι ότι μπορούμε να μάθουμε και από τα λάθη μας. Και νομίζω ότι το ΕΚΟΦΗΝ μπορεί να το κάνει αυτό, ακριβώς αυτό. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλό καινούριο χρόνο και ελπίζω αυτή ε, η νοοτροπία να αποδειχθεί ότι θα κυριαρχήσει στο ΕΚΟΦΗΝ και για τις επόμενες συνεδριάσεις του και για τα επόμενα χρόνια, γιατί η Ευρώπη τα έχει ανάγκη αυτά και μάλιστα κατεπηγόντως. Διότι αλλιώς ιδεολογικοποιούνται οι αντιμετωπίσει και δεν είναι πλέον λογικές, αλλά ιδεολογικές. Ως οικονομολόγος έχω εμπιστοσύνη στα μοντέλα και βεβαίως εφόσον τα μοντέλα αποδεικνύονται σφαλμένα τότε πρέπει να τα διορθώσω και εφόσον δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αν δεν, μπορώ, τα διορθώσω, τότε πολιτικά πανάσχημα τα πράγματα. Ο Υπουργό, σα ευχαριστώ. Αντεύχομαι για τα Χριστούγεννα και σε εσά και σε όλε και όλου του Ευρωβουλευτέ. Θα έπρεπε όμω να σα είχα, να σας είχα ευχαριστήσει ιδιαίτερω για τα ιδιαίτερα ευγενικά σα σχόλια για την πρόοδο τη Προεδρία μα, τα οποία σημειώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και θέλω να σας ευχαριστήσω και για την απάντηση που δώσατε στην ερώτηση της Ελίσας. Όντως είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και είναι δύσκολο να είναι αποτελεσματικά τα μοντέλα. Όταν όμως οι απαντήσεις είναι εσφαλμένες, δεν πρέπει να υποκρινόμαστε ότι συνεχίζουν τα μοντέλα να είναι λειτουργικά και επιτυχημένα. Ο κύριος Σμιτ τώρα για την Άλτε. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, εκ μέρου των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την φιλόδοξη Προεδρία των ε, έξι αυτών μηνών. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να ξεκινήσουν ε, κάπως ε, λανθασμένα, αλλά να έχουν τελικά μια επιτυχημένη έκβαση. Να ξεκινήσω την παρέμβασή μου παρουσιάζοντας αυτά που πιστεύω ότι δεν έχουν γίνει ακόμη. Εγώ είμαι αρμόδιος για την οδηγία για τις ε, επενδύσεις και τις ε, αποζημιώσεις και δεν φταίτε εσείς, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα από τότε που την ψηφίσαμε πέρσι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ίσονο σημασία στο ζήτημα αυτό. Εγώ θα διαφωνούσα όμως. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη. Επομένως χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα ενισχύει τις επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο. Πιστεύω ότι κάνατε λάθος στο, ε, στο, ε, ε, στο ΕΚΟΦΗΝ ως προς το θέμα της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ισορροπία δηλαδή μεταξύ των φίλων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν είναι κάτι που θα σας στοιχιώνει αλλά ενδεχομένως να στοιχιώσει, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, την ε, λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ξέρω ότι δεν φέρετε, ξέρω ότι δεν φέρετε καμία ευθύνη γι' αυτό αλλά θα ήθελα εν πάση να το δηλώσω εδώ. Έχω τρία ερωτήματα ο κύριος Κλάους Ρέγκλιν, γραμματέας του ESM, σε συνέντευξη που έδωσε χθε σε γερμανική εφημερίδα, χθε ή σήμερα, δήλωσε ότι η κρίση θα ξεπεραστεί σε δύο-τρία χρόνια και ότι οι χώρες θα επανέλθουν σε τροχιά σε δύο χρόνια, τρία, κάτι τέτοιο. Είναι μάλλον ε, αισιόδοξη αυτή η πρόβλεψη, έτσι δεν είναι. Ακούγοντας εσάς μπορεί κανείς να είναι λιγότερο αισιόδοξο βάσει το δικό σας λεγόμενο. Γιατί ήταν τόσο αισιόδοξο ο Κλάους. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, ως προς τον SSM, τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Έχουμε κάποιες χώρες που είναι πλήρως μέλη, κάποιες ε, ενδιαμέσως και κάποιες που έχουν επιλέξει να μην συμμετάσχουν. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό καταρχάς είναι καλό, καταρχήν μάλλον είναι καλό, αλλά ίσως θα μπορούσε να το ερμηνεύσει ως ε, την αρχή ε, μίας ατραπού, ε, ενός δρόμου που θα οδηγήσει σε περαιτέρω διέρεση στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας σχολιάσετε για τις πραγματικές συζητήσεις που διημήφθησαν σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ ε, φάνηκαν τα θέματα αυτά στη συζήτηση που έγινε, ακούστηκαν καθόλου. Ε, για μένα δεν είναι μόνο η Τραπεζική Ένωση, είναι ένα βήμα για κάτι άλλο στην Ευρώπη. Αυτό είναι το δεύτερο μου ερώτημα. Και το τρίτο ερώτημά μου, η Λετωνία. Έχει συζητηθεί να προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ η Λετωνία από 1η Πρώτου του 2014. Ε, ποιες είναι οι εξελίξεις ως προς το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Να διευκρινίσω, να διευκρινίσω στον Υπουργό ότι είστε ε, εισηγητής για την... Ε, για το investment compensation, το οποίο έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Εμείς το έχουμε ψηφίσει στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν έχει προχωρήσει στο Συμβούλιο νομίζω και αυτό θέλω να το διευκρινίσω. Ε, έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσω απαντώντας αντίστροφα. Ε, να ξεκινήσω απαντώντας ως προς τη Λετωνία. Εξ όσων γνωρίζω, σε επίπεδο εκοφήν δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το κατά πόσο η Λετωνία θα προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ δεν έχει συζητηθεί σε επίπεδο εκοφήν, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της εξάμενης προεδρίας μας. Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή εδώ. Τώρα, ως προς την κατάσταση ε, που έχει να κάνει με τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό και για το ποιος είναι μέσα και ποιος είναι έξω από αυτόν. Πρέπει να πω τα εξής. Πράγματι, ε, είναι ένα θέμα λεπτό και πρέπει να πετύχουμε μια λεπτή ισορροπία. Ο, ο ανιός εποπτικός μηχανικός δεν είναι για αυτούς που συμμετέχουν ή για αυτούς που δεν συμμετέχουν, είναι για όλους. Ναι. Έχει βρεθεί αυτό το ε, σύστημα και είναι ένας ενιαίος επιποπτικός μηχανισμός ο οποίος πρέπει να λειτουργήσει για όλους όσοι βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ και όλους όσοι βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ. Μέχρι αυτού του σημείου πιστεύω ότι η ισορροπία και ο μηχανισμός για τον οποίο έχει γίνει λόγος σε γενικές γραμμές ε, θα ικανοποιήσουν και τους μεν και τους δε. Εξού και μετά από μαραθώνιες συζητήσεις συμφωνήθηκε ότι πράγματι είναι εφικτός ένας τέτοιος μηχανισμός, μπορεί να γίνει, ωστόσο ε, πρέπει να ε, δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλυψε όλους αυτούς τους τομείς και περιλαμβάνει και τις δικλείδες ασφαλείας που είναι απαραίτητες για όλους. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερα να γίνουν ώστε ε, να ρυθμιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι υπήρξε καλή βούληση στη συνεδριάσεις του ΕΚΟΦΗΝ. καλή βούληση θα συνεχίσει να υπάρξει και δεν θα έχουμε διαφορετικές εκβάσεις τελικά. Θα εξευρεθούν ικανοποιητικές λύσεις πιστεύω. Και με αυτό έρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα για τα σχόλια του Κλάους Ρέκλιν ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ε, πολύ σκεπτόμενος, πολύ ικανός. Ε, σέβομαι την αισιοδοξία του ε, και μου αρέσει να πιστεύω ότι ναι, ξέρει πολύ περισσότερα από ότι πολλοί από εμά, επομένως και εγώ μοιράζομαι την αισιοδοξία του. Ίσως χρειαστούν δύο με τρία χρόνια για να ε, ανακάμψουμε. Ωστόσο, Ε, η περίοδος που έχουμε διανύσει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια κατά πάσα πιθανότητα θα καταγραφεί στην ιστορία ως μία από τις πιο τραχώδεις περιόδους της οικονομικής ιστορίας της ανθρωπότητας, η οποία δυστυχώς ε, οδήγησε σε άλλες ατυχείς και δυστυχείς κοινωνικές ε, ανισορροπίες. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση για την οποία μιλούσε ο Κλάους Ρέκλιν. Και εγώ νομίζω ότι ε, υπάρχει φως, φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Η Ευρώπη δουλεύει σταθερά για να επιλύσει όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν. Ίσως κάποια μέρα άλλες ήπειροι του κόσμου θα εξετάσουν αυτά που έχει κάνει και που κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει με αυτές τις ανεπάρκειες του συστήματος, με αυτά τα προβλήματα και θα αντιγράψουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος στον τομέα αυτό και ενδεχομένως ο Κλάους Ρέγκλιν να αναφέρεται τότε από τους ιστορικούς της εποχής ως ο άνθρωπος που ήταν πρωτοπόρος για την εξέβρεση των λύσεων και ο άνθρωπος που ήταν ο πρώτος που προέβλεψε και το τέλος αυτής της ταραχώδους ε, περίοδου. Ως προς το πρώτο σας θέμα για την προστασία των ε, επενδυτών και το σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών είναι κάτι που συνδέεται με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων βεβαίως. Και βεβαίως αυτό σχετίζεται και με το φάκελο για τη διαχείριση ε, των κρίσεων, τον οποίο εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε πρόοδο πρώτα ε, στα θέματα της διαχείρισης της κρίσης για να μπορέσουν να υπάρξουν και εξελίξεις ε, σε σχέση με την οδηγία αυτή για την αποζημίωση των επενδυτών. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ εκ μέρους του ΕΛΚ, κυρία Ρόδη Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Υπουργέ, ε, σε συνέχεια αυτό που ήδη εσείς έχετε αναφέρει και οι συνάδελφοι ρώτησαν, ε, ήθελα να σας απευθύνω κι εγώ μια σχετική ερώτηση που έχει να κάνει με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. απαντήσετε άμεσα ή έμεσα για τα, τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από την, ε, το καλό σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών, την επιτυχή ε, εφαρμογή τους. Αυτό που θα σας ρωτήσω, υπάρχουν συζητείτε στο ΕΚΟΦΗΝ για συμπεράσματα που μπορεί να είναι χρήσιμα ε, σε άλλες χώρες όπως παραδείγματος χάρη Κύπρος τώρα που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Γίνεται λόγος δηλαδή για προσαρμογές λαμβανωμένων υπόψη των, ε, των συμπερασμάτων. Και το άλλο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι σχετικά με την ε, εναρμόνιση φορολογίας. Ε, έχει η Κυπριακή Προεδρία ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, έχει κάτι να μας επισημάνει. Βλέπουμε ότι από τη μια μεριά υπάρχει ανάγκη συντονισμού της φορολογίας, από την άλλη μεριά είναι ένας μοχλός για την ανάπτυξη. Βλέπουμε η Πορτογαλία τώρα που ζητάει από την Τρόικα να διευκολυνθεί με 10% φορολογία στις νεοσύστατες της επιχειρήσεις για να ε, ε, συμβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας της. Έχετε κάτι να σχολιάσετε από αυτού. Ευχαριστώ. At level. Σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ δεν συζητούμε τέτοιες λεπτομέρειες, ειδικότερα όσον αφορά στη φορολόγηση και μάλιστα σε συγκεκριμένες χώρες. Τα βασικά ζητήματα που συζητούνται σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ, όπως καταλαβαίνετε, είναι πώς μπορεί να δοθεί βοήθεια στις χώρες που ε, μπαίνουν σε πρόγραμμα ε, δημοσιονομικής προσαρμογής. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, το πρόγραμμα υποβλήθηκε πριν από αρκετό καιρό, γίνονται ε, τριμηνιές αναθεωρήσεις και εκεί ε, μετράται η πρόοδος, γίνονται προσαρμογές στο πρόγραμμα, προσφέρονται χαλαρώσεις όπου δει, ζητούνται επιπρόσθετα μέτρα όπου δει, αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο σε επίπεδο τρόικας και έρχονται στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ προς έγκριση. Το ΕΚΟΦΗΝ δεν θα ξεκινήσει από μόνο του να θέτει ε, θέματα όπως αυτά που αναφέρατε, για παράδειγμα θέματα φορολογίας. Και σε κάθε περίπτωση στην, ως προς την Κύπρο η οποία βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας και ε, συμφωνίας επί ε, μνημονίου κατανόησης το οποίο έχει τύχει η συμφωνία στο μεγαλύτερο μέρος του ένα σημειωμένη εκρεμές δεν έχει ολοκληρωθεί γι' αυτό περιμένουμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων στην περίπτωση της Κύπρου δεν έχουν τεθεί τέτοια θέματα σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ε, Ρεϊνάλτο Ντομινίτσι, εξ ονόματος των ε, Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάω Ιταλικά. Πιστεύω πως, όπως είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι η εμπειρία των οργανισμών αξιολόγησης ήταν ε, μια σημαντική στιγμή, ένα ορόσημο για τις εργασίες της Κυπριακής Προεδρίας. Υπήρξαν σημεία δυσκολίας που εν μέρη ξεπεράστηκαν. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, ούτε για το περιεχόμενο της συμφωνίας που τελικά επετεύχθη μετά από μακρές και κουραστικές διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα σύντομα να κάνω ένα σχόλιο για τον τρόπο εργασίας του Συμβουλίου, τη λειτουργία του και το ρόλο του και να σας θέσω ένα ερώτημα καθώς και να προτείνω κάτι. Και την πρόταση την κάνω αμέσως. Με βάση την εμπειρία των διαπραγματεύσεων για τις, ε, ε, τους οργανισμούς αξιολόγησης θα μπορούσε η Κυπριακή Προεδρία να αφήσει στους διαδόχους της και εν γέννη στο Συμβούλιο έναν κρίσιμο ε, προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η εμπειρία εργασίας συνέχισε. Δηλαδή, Καταρχήν, από αυτό που πριν ε, εργαζόταν το Συμβούλιο, να μια κάποια έλλειψη διαφάνειας, μια κάποια αδιαφάνεια. Μια ερώτηση για την διαβίβαση της πολιτικής βούλησης εντός του Συμβουλίου. Δηλαδή, ποιος αποφασίζει τις αποφάσεις που θα ληφθούν και ποια στάση θα διατηρηθεί απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα, ξεκινώντας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμπειρογνώμονες, διπλωμάτες, εκπρόσωποι των ε, κυβερνήσεων. Έπειτα ένα πρόβλημα εξωτερικής επικοινωνίας ε, συμβαίνει, δεν με ακούτε καλά, μήπως. Υπάρχει πρόβλημα με την ε, μετάφραση. Ρωτάει ο κύριος Δομέντσι. Μ' ακούτε καλά. Λοιπόν, ένα πρόβλημα που εν γέννη αφορά την δυνατότητα να διεξάγονται καλύτερα και πιο με μεγαλύτερη διαφάνεια εργασίες ε, του Συμβουλίου επί τη βάση αυτής της ειδικής συγκεκριμένης εμπειρίας και τις συγκεκριμένες διαπραγμάτευσεις για, τις, ε, για τους οργανισμούς ε, αξιολόγησης. Εγώ έχω ριζοσπαστική άποψη για την, ε, το Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω πως το Συμβούλιο είναι το βασικό εμπόδιο στο δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να θέσω αυτό το ζήτημα της λειτουργίας του με βάση τη συγκεκριμένη εμπειρία. Δεύτερο ερώτημα αφορά την ουσία, το περιεχόμενο των θέσεων για τις, ε, τους οργανισμούς πιστοληπτικής ε, ε, αξιολόγησης. Όταν εγώ συναντήθηκα με τον πρέσβη Κορνελίου, το ίδιο ερώτημα είχαμε εγώ και εκείνος. Γιατί για το συγκεκριμένο θέμα για τους οργανισμούς αξιολόγησης ήταν τόσο δύσκολο να συνεργαστούμε με τους ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεδομένου ότι αυτές οι ίδιες κυβερνήσεις σε ορισμένες ε, εμφάσεις έδειξαν ε, πολύ μεγάλες, ε, μάλλον άσκησαν δρυμία κριτική απέναντι σε αυτές τις οργανισμούς. Αλλά τη στιγμή της λήψης σημαντικών αποφάσεων οι ίδιες κυβερνήσεις τράβηξαν χειρόφρενο, έκαναν πίσω και στη φάση αυτή είχαμε σημαντική δυσκολία για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Με βάση λοιπόν αυτή την εμπειρία τη συγκεκριμένη σας ρωτώ, η Κυπριακή Προεδρία μπορεί να αφήσει ένα είδους ε, κληροδοτήματος στις επερχόμενες προεδρίες ώστε να διορθωθούν κάποια προβλήματα στον τρόπο εργασίας του Συμβουλίου και για το συγκεκριμένο πρόβλημα των οργανισμών αξιολόγησης. Ευχαριστώ. Um, I um, uh, Γνωρίζω την άποψη αυτή και πιο συγκεκριμένα την ε, προσωπική σας γνώμη όσον αφορά την, τον ρόλο του Συμβουλίου. Βεβαίω θα κατανοήσετε ότι η Προεδρία παίρνει την εντολή της από τα κρατημέλη Και οι διπλωμάτες από τις κυβερνήσεις τους. Άρα λοιπόν η Προεδρία είναι απλά ο συντονιστής ανάμεσα στα κρατημέλη. Εάν η ερώτηση που θέσατε είναι κατά κάποιο τρόπο η δημοκρατική νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τότε η απάντησή μου θα ήταν ότι είμαστε πεπισμένοι ότι οι ισχυροί μηχανισμοί δημοκρατικής νομιμότητας είναι απαραίτητοι. Στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου συμφωνήθηκε ότι τα κράτη-μέλη θα εμπλέκουν καταλήλως τα εθνικά τους κοινοβούλια όταν και όσον αφορά την περαιτέρω ολοκλήρωση των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών τους. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της συνθήκης, της συνθήκης ε, περί σταθερότητας, συντονισμού και διακυβέρνησης, η περιβάση του πρωτοκόλλου παριθμών 1, η συνεργασία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό θα ενισχυθεί Άρα λοιπόν εξαρτάται από τα εθνικά κοινοβούλια και από το, και από το ευρωπαϊκό να καθορίσουν πώς θα οργανώσουν την επικοινωνία μεταξύ τους για να συζητούν αυτά τα θέματα όπως ας πούμε το Ιωνέ. Πολλά ακόμα βεβαίως θα πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί αυτή η δημοκρατική νομιμοποίηση. Αλλά σέβομαι τις προσωπικές σας απόψεις σχετικά με το Συμβούλιο. Thank you. Um, ευχαριστώ. Δεν έχω κάποιον άλλο μιλητή από το ΕΛΚ αυτή τη στιγμή. Όχι. Οπότε, εξ ονόματος των σοσιαλιστών, Ιάννη Ποδηματά. Uh, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, ε, μπορείτε να μου απαντήσετε αγγλικά, αλλά επειδή σπανίως έχουμε ελληνική προεδρία, ελληνόφωνη προεδρία του Συμβουλίου, θέλω να σας μιλήσω στα ελληνικά. γιατί, και να σας συγχαρώ για την εξάμεινη προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ε, και για το ρόλο που αποδώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γιατί προχωρήσατε πολύ σημαντικούς φακέλους ε, για μας, για την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ιδιαίτερα θέλω να σας ευχαριστήσω ως εισηγήτρια της έκθεσης για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, διότι παρά τις ε, διαφωνίες μας επί της ουσίας της πρότασης, η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργήσε ως ε, έντιμος διαμεσολαβητής και προχώρησε το φάκελο με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε στη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας. Με αφορμή ωστόσο αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ, θέλω να επιμείνω στα θέματα της φορολογίας. Νομίζω ότι η συνάδελφος Ρόδη Κράτσα έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι η φορολογία είναι ένα εργαλείο ε, που μπορεί να παίξει καταλητικό ρόλο, ε, μπορεί να είναι αιχμή του δόρατος για μια κοινωνικά δίκαιη αλλά και φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε τη θέση ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς ένα περισσότερο ενιαίο πλαίσιο στα θέματα της φορολογίας, με δεδομένο ότι η βαθύτερη δημοσιονομική ολοκλήρωση πηγαίνει χέρι-χέρι με την φορολογική εναρμόνιση και αν συμφωνείτε να αποδοθεί δεσμευτικός χαρακτήρας στο σχέδιο της Επιτροπής για την πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και για την κοινή φορολογική βάση και την οδηγία φορολόγησης καταθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για τα πολύ ευγενικά σας σχόλια για την Προεδρία μας και για τη δουλειά που κάναμε. Πρέπει να πω ότι ναι, η Κύπρος είναι με μικρή χώρα, αλλά ανέλαβε αυτό το καθήκον ε, με επιφυλάξεις. Αναρωτιόμασταν αν θα ήμασταν έτοιμοι και θα μπορούσαμε να τα φέρουμε σε πέρας όλα αυτά. Από αυτή τη διαδικασία όμως μάθαμε το εξής εάν συγκεντρώνεται κανείς ε, στο σκοπό του και αν πιστεύει στην Ευρώπη και αν βασιστεί στη βοήθεια των κρατών μελών, την οποία πράγματι είχαμε, τότε μπορούμε να πετύχουμε πολλά ε, στην Προεδρία μας, όσο και οποιαδήποτε άλλη χώρα, παρόλο που μπορεί να είναι πιο μεγάλη. Και αυτό είναι ένα ε, μάθημα που μάθαμε αυτούς τους έξι μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας λόγια, λοιπόν. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο το οποίο σκέφτηκα μετά την ερώτηση του κυρίου Γκοζές. Ένα από τα ε, πράγματα που μάθαμε κατά τη διάρκεια της εξάμενης προεδρίας μας είναι το εξής. Ε, έφερε το λαό μας πιο κοντά στην Ευρώπη η προεδρία αυτή και αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Εάν ε, πρόκειται να είμαστε Ευρωπαίοι, τότε πράγματι πρέπει να έχουμε μια κοινή βάση, να πιστεύουμε σε κάποιες κοινέ αξίες. Και η Κυπριακή Προεδρία ήταν ευκαιρία για μας προς αυτή την κατεύθυνση. Κοινέ αξίες ώστε να καταλάβουν όλοι περί τίνος πρόκειται. Η εμπλοκή μας στην Προεδρία κατά τη διάρκεια των έξι αυτών μηνών ήταν αρκετή για να πιστέψουμε και να ενστερνιστούμε αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες πολύ περισσότερο από ό,τι, το είχαμε κάνει στο παρελθόν ή από ό,τι θα το κάναμε ποτέ ούτως ή άλλως. Ε, και έρχομαι τώρα στο θέμα των κοινών αξιών και των κοινών προσεγγίσεων. Μία κοινή προσέγγιση στη φορολογία, για παράδειγμα, είναι κάτι ε, που μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα επιβάλλοντας έναν π.χ. φορολογικό συντελεστή παντού. Η έμεση φορολογία είναι ήδη ενερμανισμένη. Χρειάζεται ομοφωνία, όπως γνωρίζετε, ε, στα φορολογικά για να αλλάξει οτιδήποτε. Αλλά μια κοινή βάση, ναι, μπορεί να επιτευχθεί και πρέπει να εξεταστεί ε, στο πλαίσιο των διαφορετικών χωρών, των διαφορετικών οικονομιών. Διότι δεν είναι αυτός ο μόνος παράγοντας που καθορίζει τις οικονομικές εξελίξεις και την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Δεν είναι η φορολογία αυτή που ε, καθορίζει την οικονομική μοίρα μιας χώρας μόνο. Ε, πρέπει να εναρμονίσουμε όσο το περισσότερο αυτό ναι και έχει γίνει αυτή η δουλειά τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά ακόμα προφανώς, λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες κάθε χώρας. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, σε όλα τα άλλα ζητήματα. Ε, να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση ε, ως προς τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό υιοθετήθηκε, αποφασίστηκε την περασμένη εβδομάδα, προστατεύοντας όμως τα συμφέροντα όλων, είτε θα ε, είναι μέσα είτε θα είναι έξω από αυτό το μηχανισμό. Χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα προφανώς, αλλά οι κοινέ αρχές θα πρέπει να ισχύσουν ακόμα και στην, ε, στον τομέα της φορολόγησης. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ εξ ονόματος των σοσιαλιστών, ο Αντολίν, Ζητώ συγγνώμη διότι δεν παρακολούθησα την αρχική σας παρέμβαση γιατί ήμουν στην Επιτροπή αλληλία, διότι συζητείται εκεί η έκθεση για την οποία είμαι εισηγητής και γι' αυτό ήρθα καθυστερημένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ για τη συνεργασία ε, που είχατε ως προς την νομοθετική πρωτοβουλία ε, για την μεταρρύθμιση ε, των υποθηκών και των ε, δανείων. Ελπίζω ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα συνεχίσει να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μοιραστείτε με τους Ιρλανδούς συναδέλφους ε, την ανησυχία μας. Πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό το φάκελο ώστε να μην υπάρξουν τέτοια προβλήματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν στις χώρες σε όλο αυτό τον κλάδο των δανείων. Κάτι το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Ο Υπουργό σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Πράγματι, αναλαμβάνω αυτή την υποχρέωση. Θα μεταβιβάσω το μήνυμά σας ε, στην νέα την επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία. Ε, γνωρίζω πόση σημασία δίδεται στο ε, θέμα αυτό και καλώς βεβαίως το κάνετε η Πρόεδρος, ε, έχουμε εξαντλήσει τον κατάλογο των ομιλητών. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο αυθόρμητα τώρα. Η Ελίσσα παρακαλώ. Δεδομένου ότι έχω την ευκαιρία να θέσω ερώτημα, κυρία Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να πω το εξή. Ω προ τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, έχω κάποια λεπτομερή ερωτήματα να θέσω. Δεν ξέρω αν εσεί είστε αρμόδιο να μου απαντήσετε, αλλά προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώ ακριβώ θα λειτουργήσει αυτό ο μηχανισμό. Επομένω, πρόσβαση υπάρχει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και συνδέεται αυτό με την άμεση χρηματοδότηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών και αυτό θα γίνει μετά που θα ε, μπουν οι τράπεζες στην εποπτεία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Τώρα όμως έχουμε τράπεζες οι οποίες ε, είναι άμεσα υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχουμε και άλλες τράπεζες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών. Οι τράπεζες που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ε, financial backstop σε σχέση με αυτές που εποπτεύονται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή θα υπάρξει διαχωρισμός στην πρόσβαση αναλόγως με το είδος των τραπεζών. Δεν ξέρω αν καταλάβατε το ερώτημά μου. για το θέμα του backstop ως κριτήριο. Μπορείτε να το επαναλάβετε, λέει ο κ. Υπουργό. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε ε, τράπεζες που έχουν συστημική σημασία και είναι υπό τον άμεσο έλεγχο, υπό την άμεση εποπτεία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτές που έχουν ε, συστημική σημασία, ε, αυτό είναι το κριτήριο που έχει εδρεωθεί, ε, κάποιες τράπεζες είναι υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 130 ε, περίπου τράπεζες, έτσι δεν είναι. Ο κύριος Υπουργός, να διευκρινίσω το εξής. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εποπτεύει άμεσα καμία τράπεζα, κανενός, κανενός μεγέθους. Μιλούμε για το τι προτίθεται και τι προτείνεται να γίνει τους επόμενους μήνες. Μιλούμε για ένα σύστημα το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από το 2014. Ναι, τα γνωρίζω αυτά, λέει η κυρία Φερέιρα. Καλώς. Ε, έκανα λάθος το χρόνο του ρήματος. Εν πάση περιπτώσει, προβλέπετε οι τράπεζες, είτε εάν πρόκειται να είναι υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε αν πρόκειται να είναι υπό την εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών, θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δυνατότητες άμεσης ανακεφαλοποίησης από το ε, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή θα έχουν ε, ανακεφαλοποίηση από διαφορετικές πηγές. Ο Υπουργός. Νομίζω ότι έχετε πάει πολύ πιο πέρα από ό,τι έχουμε ήδη συζητήσει. Θέλω να σας εξηγήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να εποπτεύει όποια τράπεζα επιλέξει η ίδια, χρησιμοποιώντας κριτήρια. Ε, υπάρχουν ήδη κάποια κριτήρια για το ποιες τράπεζες θα εποπτευθούν. Καταρχάς οι μεγαλύτερες τράπεζες, γιατί έχουν καθοριστεί τα κριτήρια, ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή η Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει όσο περισσότερες τράπεζες μπορεί να διαχειριστεί, να αναλάβει την εποπτεία τους εννοείται. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα αυτό και στην πράξη δεν θα εποπτεύσει άμεσα 6.000 τράπεζες π.χ. Αυτή τη στιγμή περιορίζει το αριθμό των τραπεζών που θα εποπτεύσει άμεσα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, όταν τίθεται και αν τεθεί το θέμα της άμεσης ανακεφαλοποίησης μιας τράπεζας, τότε το ζήτημα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και να εξεταστεί αναλόγως με τη χρονική συγκυρία, τις ειδικέ περιπτώσεις, τις ειδικέ συνθήκες που αφορούν την εκάστοτε περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Η απόφαση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή αφήνει την πόρτα ανοιχτή ώστε να υπάρξουν ειδικέ εξαιρέσεις που μπορούν να εξεταστούν και νωρίτερα, πριν από το 2014, όποτε θα αρχίσει να ισχύει και όλας ο νέος εποπτικός μηχανισμός. Ε, πρέπει να είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις και να τεθούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Πρόεδρος. Νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε να διευκρινιστεί το ζήτημα αυτό στον, τριμερο, στον τριμερή διάλογο, ο οποίος θα ξεκινήσει αύριο. Όλα περιλαμβάνονται στον ενίο εποπτικό μηχανισμό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το δικαίωμα παρέμβασης. Ενδεχομένως θα πρέπει μετά να αναλάβει μια τράπεζα της οποίας η εποπτεία αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη. Θα τα δούμε αυτά. Ε, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά όταν ε, ήρθα για πρώτη φορά να σας δω στην Κύπρο, θυμάμαι ότι είχατε δεχθεί να αναλάβετε το ρόλο αυτό λόγω της ε, τεχνικής σας ε, κατάρτισης διότι δεν προέργεστε άμεσα από το κόσμο της πολιτικής και μου είχατε πει ότι ναι, αναλαμβάνω το αξίωμα αυτό για να βοηθήσω εγχωρίως την κατάσταση. Νομίζω ότι ε, αναλάβατε πάρα πολλά βάρη, πολύ περισσότερο από ό,τι είχατε υπολογίσει εξ αρχής και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, διότι πιστεύω ότι ε, είχατε μία αναζωογονητική ειλικρίνεια στις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις και αυτό συνοδεύεται από τη βαθιά σας ε, ε, τεχνική ε, κατάρτιση. Σας εύχομαι τώρα καλή ξεκούραση. Σας συγχαίρω για όλα αυτά τα οποία καταφέρατε και για τις μαραθώνιες συζητήσεις για το δανείο εποπτικό μηχανισμό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Να έχετε καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Αύριο το πρωί να πω ότι θα συνεδριάσουμε στην αίθουσα 2Q2, όχι εδώ, στις 9 ακριβώς. Ευχαριστώ όλους.